Uh, Συνάδελφοι, καλημέρα. Ας ξεκινήσουμε με το θέμα υπαριθμών 13, κατάσταση προόδου των εμπορικών διαπραγματεύσεων με το Μεξικό. Λοιπόν, στις 9 Νοεμβρίου είχαμε την τελευταία συζήτηση εδώ στην Επιτροπή για το θέμα αυτό και έγινε και μια επίσημη αποστολή στο Μεξικό το 2017. Οι διαπραγματευτέ είχαν θέσει φιλόδοξη προθεσμία για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων έως το τέλος του 2017. Αυτός ήταν ο στόχος, κατά την, ε, να υπάρξει η ολοκλήρωση αυτή κατά την υπουργική διάσκεψη του ΠΟΕ. Δυστυχώς όμως αυτό φαίνεται να μην κατέστη δυνατό. Συνεχίζονται λοιπόν οι διαπραγματεύσεις και θα θέλαμε να μάθουμε σήμερα σε ποιο σημείο βρισκόμαστε. Έχουμε μαζί μας σήμερα εδώ εκπροσώπους της ε, Μεξικανικής Πρεσβείας. Σας καλωσορίζω. Και την επικεφαλής των διαπραγματευτών της ε, Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου, την κυρία Έλενα Κούνιχ. Θα ήθελα να δώσω το λόγο πρώτα στην κυρία Κόνιχ, στη συνέχεια να δώσω το λόγο στην κυρία Ροντρίγε Πινιέρο, που είναι η συγγήτριά μας για το Μεξικό, και στη συνέχεια στα μέλη της Επιτροπής. Κυρία Κόνιχ, παρακαλώ πείτε μας που βρισκόμαστε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, με χαρά είμαι εδώ. Όπως είπε και ο πρόεδρος, είχαμε ένα φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα, ελπίζοντας ότι θα μπορούσαμε να κλείσουμε τις διαπραγματεύσεις μέχρι το τέλος του 2017. Τώρα και οι δύο πλευρές συμφωνούν ότι αυτός ήταν ένας πολύ φιλόδοξος στόχος. Το πιο σημαντικό όμως είναι, είναι ότι και οι δύο πλευρές θα φτάσουν σε μια συμφωνία υψηλού επίπεδου που θα είναι επωφελής και για τις δύο πλευρές και τις οικονομίες τους. Έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδο στο γύρο διαπραγματεύσεων τον Δεκέμβριο. Υπάρχουν διάφορα θέματα εκκρεμή. Πολλά θέματα επιλήθηκαν. Αλλά υπάρχουν ακόμα και θέματα κλειδιά που δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Δεν είναι ασύνηθες αυτό ε, σε τέτοιου τύπου διαπραγματεύσεις ε, μεταξύ της της 12 και 21 Δεκεμβρίου στο, στην πόλη του Μεξικού ε, συμφωνήσαμε 8 κεφάλαια, εμβαθύναμε τις συζητήσεις σε κάποια από, βασικά, τα βασικά εκκρεμή θέματα που πρέπει να επιληθούν για τις ε, δημόσιες συμβάσεις, όπου ένα από τα βασικά δικά μας θέματα είναι να καλύψουμε το υπομοσπονδιακό επίπεδο γιατί υπάρχει σημαντική κάλυψη σε ομοσπονδιακό επίπεδο ή στην ισχύου συμφωνία του 2000. Κάναμε επίσης καλές συζητήσεις για τις υπηρεσίες. Υπάρχουν ανοιχτά θέματα για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, ε, για την προσωρινή απομάκρυση ε, ανθρώπων Mode 4, θέματα δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, κυρίως κανονιστική προστασία δεδομένων, διπλώματα ευρεσιτεχνία δηλαδή. Κάναμε καλή πρόοδο για νέα κεφάλαια, καταπολέμηση διαφθοράς, δηλαδή. Σημαντική πρόοδο για τις υπηρεσίες γενικότερα, όπου ανταλλάξαμε προσφορές. Επίσης, Έχουμε καλές αλλά προβληματικές συζητήσεις ε, για τις γεωγραφικές ενδείξεις. Δεν είναι περίεργο. Είναι σημαντικό ενδιαφέρον για την Ευρωπαϊκή Ένωση και φυσικά υπάρχουν ε, μεξικανικές βιομηχανίες που θέλουν να παραμείνουν τα αγαθά τους ε, στην αγορά. Ορισμένα από αυτά τα αγαθά είναι στη μεξικανική αγορά επί μακρόν. Επίσης κάναμε συζητήσεις για την τελευταία προσφορά για την πρόσβαση στην αγορά αγαθών και λογικό είναι ότι θα γίνουν περαιτέρω συζητήσεις για το θέμα αυτό καθώς μπαίνουμε στην τελική φάση. Από το γύρο διαπραγματεύσεων στην πόλη του Μεξικού τέλη του 2017 ε, ήρθαμε σε επαφή μετά αφού τελείωσε επανήλθαμε, ήμασταν σε επαφή οι δύο διαπραγματεύτικέ ομάδες. Την, προηγούμενη, την προπροηγούμενη εβδομάδα είχαμε επαφές και θα έρθουμε... Θα έρθει η Μεξικανική ομάδα στις 5 Φεβρουαρίου αυτή τη εβδομάδα. Και εμείς θα πάμε στην την ε, εβδομάδα, που, Δευτέρα δηλαδή 12 και όλη τη εβδομάδα. Έντονες συζητήσεις θα πρέπει να υπάρξει σημαντική δέσμευση για να κλείσουν αυτές τις διαπραγματεύσεις το δυνατότερο αρχές του 18 θα θέλαμε εμείς, παρότι δεν έχουμε θέσει οριστική ημερομηνία. Θα θέλαμε να κλείσουμε πάντως πριν τις εκλογές και την προεκλογική εκστρατεία στην πόλη του Μεξικού. Το Μεξικό έχει ε, προεδρικές και κοινοβουλευτικές εκλογές 1η Ιουλίου. Και 1η Μαρτίου ξεκινά επίσημα η προεκλογική εκστρατεία. Οι ομάδες θα συναντηθούν, θα έχουμε και υπουργικές επαφές και ελπίζουμε ότι ο Επίτροπος Γουαχάρο και η Επίτροπος Μάρτρομ θα συναντηθούν στις Βρυξέλλες αυτή τη βδομάδα. Η, η κυρία Μάρτρομ είναι έτοιμη να πάει στην πόλη του Μεξικού μια και είμαστε στην τελική φάση των διαπραγματεύσεων, αλλά θα πάει όταν ε, θα έχουν ε, ουσιαστικά ε, λυθεί τα θέματα και θα έχουν παραμείνει ένα-δύο θέματα κλειδιά, ας που θα πρέπει να επιληθούν σε υπουργικό επίπεδο. Βασικό κλειδί για να έχουμε καλά αποτελέσματα στη διαπραγμάτευση είναι να έχουμε μια μοντέρνα εκδοχή της παλιάς συμφωνίας. Το ξαναείπα αυτό. Η παλιά συμφωνία είναι σε ισχύ εδώ και 15 χρόνια. Έχουν γίνει αλλαγές στο μεταξύ στο Μεξικό, στην νομοθεσία του και από πλευράς μας έχουν γίνει αλλαγές μέσα αυτά τα 15 χρόνια. Και φυσικά όταν έχεις ήδη μια συμφωνία υπάρχουν λιγότερα πράγματα που πρέπει να επιληθούν. Παρ' όλα αυτά σε όλα τα κεφάλαια σχεδόν πρέπει να υπάρξουν επικαιροποίησεις. Όσοι ξέρουν τη συμφωνία και την, έχουν διατρέξει την, το που έχουμε φτάσει ε, το Δεκέμβριο θα το ξέρουν αυτό. Επίσης ε, για την πρόσβαση στην αγορά υπάρχουν επιπλέον προσφορές και ιδίω για τα αγαθά ε, τώρα μιλάμε και για τα γεωργικά προϊόντα που δεν είχαν συμπεριληφθεί στην προηγούμενη συμφωνία. Επίσης, ε, περνάμε από το μοντέλο ISDS, ε, επίλυσης δηλαδή διαφορών μεταξύ κράτους και επενδυτών, στο, σε, σε, επίπεδο, στο μοντέλο δηλαδή δικαστηρίου για την επίλυση των διαφορών και σε υπομοσπονδιακό επίπεδο. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ πολύ και την Επιτροπή για τις εξηγήσεις που μας έδωσε. Εγώ ως εισηγήτρια εξ νόμο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις εμπορικές σχέσεις με το Μεξικό ε, θα πρέπει να τονίσω πόσο μεγάλη σημασία έχει για τους δύο εταίρους ε, η επίτευξη μιας καλής και φιλόδοξης συμφωνίας και ε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε ε, τους κοινούς μας στόχους, να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις και να μην έχουμε ε, μία συμφωνία που να μένει πίσω σε σχέση με τις συμφωνίες της υπόλοιπης που έχουμε υπογράψει. Και γι' αυτό και εκτιμώ την προσπάθεια διαπραγμάτευσης από πλευρά των δύο, του Μεξικού και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμμερίζομαι απόλυτα ότι καθώς είναι πολύ σημαντικό να επιτευχθεί η ολοκλήρωση της συμφωνίας πριν από την έναρξη της προεκλογικής εξαρτίας και να μπορέσουμε εδώ στο Κοινοβούλιο να ψηφίσουμε αυτή τη συμφωνία, είναι σημαντικό να ε, εξετάσουμε εις βάθος το περιεχόμενο. Θέλω να κάνω κάποιες ερωτήσεις ε, ώστε να Έχουμε κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες από πλευράς της Κομισιόν και των εκπροσώπων του Μεξικού, τους οποίους καλωσορίζω κιόλας με την ευκαιρία σε σχέση με τις ε, δημόσιες ε, προμήθειες. Τονίσαμε ότι υπάρχει ε, το επίπεδο κάτω από το ομοσπονδιακό, το οποίο είναι σημαντικό για μας και θα ήθελα να, να μου πείτε περισσότερα πράγματα ε, για το πού ακριβώς βρισκόμαστε και πώς σκοπεύετε να επιλύσετε το συγκεκριμένο θέμα. Τώρα, όσον αφορά την επίλυση των διαφορών, το Μεξικό, από ό,τι φαίνεται ήδη ε, έχει δεχθεί την πρόταση το Μεξικό. Όμως, Ποια θα ήταν η θέση του Μεξικού σε σχέση με την ευρωπαϊκή πρόταση να δημιουργηθεί ένα πολυμερές δικαστήριο, δηλαδή έτσι ώστε όπως μάλλον και το ε, επενδυτικό δικαστήριο που είχαμε ήδη ε, συζητήσει. Τώρα, έχουμε δυσκολίες στο να έχουμε δύο διαφορετικά συστήματα. Το μεξικανικό σύστημα επικεντρώνεται στα σήματα και το δικό μας ε, σύστημα ε, στη γεωγραφική ε, προέλευση έχει διαφορετικό τύπο και στον Καναδά υπήρχε διαφορετικό πρότυπο. Το λύσαμε όμως το θέμα και λειτουργεί το σύστημα. Τι γίνεται σε σχέση με το Μεξικό όσον αφορά την βιώσιμη ανάπτυξη και με βάση τις πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί είδαμε ότι βρισκόμαστε στον 7ο γύρο διαπραγματεύσεων το Δεκέμβριο και η, η Κομισιόν είπε ότι ολοκληρώθηκε η συζήτηση για το θέμα, η διαπραγμάτευση μάλλον σε σχέση με την ε, βιώσιμη ανάπτυξη. Μας θέλω να δω πώς ολοκληρώθηκε, ποιοι είναι οι στόχοι, πού εστιάζει περισσότερο η Κομισιόν ώστε να εγγυηθεί εμπόριο και βιώσιμη ανάπτυξη με συνοχή, φιλοδοξία και αποτελεσματικότητα. Έπειτα, ποιε ε, προβλέψεις και ποιοι έλεγχοι γίνονται όσον αφορά το εργατική νομοθεσία, την περιβαλλοντική νομοθεσία ε, σε σχέση με τους ε, βασικούς κανόνες του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας και σε σχέση με τη συμφωνία που επιτέφθη στο Παρίσι και σχέση με το φύλλο τώρα. Δεν έχουμε δική συμφωνία για την ισότητα των φύλων όπως ε, στη συμφωνία με τη Χιλή. Η Κομισιόν σκέφτεται να περιλάβει τέτοιες διατάξεις όσον αφορά τα δύο φύλλα κάτι που και για το Μεξικό θα ήταν πολύ σημαντικό να ενταχθούν, δηλαδή μηχανισμοί που θα επιτρέπουν μέσω αυτής της συμφωνίας να βοηθήσουν ώστε οι γυναίκες να μπορούν να χαίρουν το διεθνούς δικαίου. Και για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εχθές είχαμε το λυπηρό νέο ε, των αποτελεσμάτων της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, το, η διάρκεια του 2017 στο Μεξικό. Πάνω από 25.000 ανθρωποκτονίες, 70 άνθρωποι διολοφονούνται την ημέρα. 1.500 ανοιχτές υποθέσεις για ανθρωποκτονία σύμφωνα με το Εθνικό ε, ε, Στατιστικό Σύστημα και υπάρχουν πολύ περισσότερες δηλαδή υποθέσεις από ό,τι το περασμένο χρόνο. Κάθε... Και φτάνουμε στις ε, ε, στα δυσθεώρητα νούμερα του πολέμου κατά των ναρκο... Ε, της, της διακίνησης ναρκωτικών, κατά των ε, αρχηγών των καρτέλ. Πώς θα καταπολεμήσετε αυτή το... αυτό το πρόβλημα. Έπειτα υπάρχουν συγκεκριμένες διατάξεις όσον αφορά το ξέπλυμα χρήματος. Πώς δεχτήκατε το Μεξικό την πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πώς έχουν προχωρήσει, ε, έχει προχωρήσει ο τελευταίος γύρος των διαπραγματεύσεων σε σχέση με αυτό το θέμα. Τώρα όσον αφορά τη διαφάνεια. Εχθές ε, Ακούσαμε και ένα ευχάριστο νέο ότι το κοινοβούλιο αυτό, αυτή εδώ η επιτροπή, η ομάδα μου διεκδίκησε επίμονα τη δημοσίευση της εντολής του Συμβουλίου όσον, όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις και χθες ανακοινώθηκε και δημοσιεύθηκε η εντολή για τη Χιλή, αλλά δεν θα πρέπει αυτό να αποτελέσει την εξαίρεση ούτε κάτι το περίεργο, θα πρέπει να είναι το στάνταρ. Θέλω να ξέρω λοιπόν πότε προβλέπετε να δημοσιεύσετε την εντολή τη διαπραγματευτική με το Μεξικό μετά από 8 γύρους διαπραγματεύσεων και σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα υπάρχει ένα θέμα που με ανησυχεί. Πότε προβλέπετε να ολοκληρωθεί η ε, μελέτη αντικτύπου και η μελέτη βιωσιμότητας και σκοπιμότητας. Θεωρείτε ότι θα καταφέρουμε Αυτή μας η επιθυμία που θεωρώ ότι είναι και ανάγκη να ψηφιστεί αυτή η συμφωνία ε, σε αυτή τη θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Τώρα οι σκιώδες εισηγητές. Πρώτα η Έμα Μακλάφριν. Ευχαριστώ Πρόεδρε, συμφωνούμε όλοι ότι αυτή η συμφωνία Μεξικού Ευρωπαϊκής Ένωση πρέπει να επικυρωθεί το συντομότερο δυνατό και γι' αυτό λόγο είναι απογοητευτικό το γεγονός ότι δεν καταφέραμε να τηρήσουμε τη δική μας προθεσμία που είχαμε θέσει για το Δεκέμβριο του 2017. Τα ερωτήματά μου λοιπόν θα κατευθυνθούν προ το γιατί δεν καταφέραμε να τηρήσουμε αυτή την προθεσμία. Πολλά θέματα ήδη τέθηκαν από την εισηγήτρια, τι δημόσιε προμήθειε, την καταπολέμηση διαφθορά και άλλα. Εγώ θεωρώ ότι ε, το Μεξικό περιμένει αυτή τη στιγμή να ακούσει τις προτάσεις της Κομισιόν. Ε, ακούσαμε πολλές φορές και έχουμε ακούσει πολλές φορές στο παρελθόν ότι υπάρχουν αυτές οι προτάσεις ε, κτλ. κτλ. Το ερώτημα είναι για ποιε είναι ακριβώ οι προτάσει που έχουν τεθεί επιτάπητο και που συζητούνται αυτή τη στιγμή μεταξύ των δύο πλευρών. Όσον αφορά την ε, συνεχιζόμενη ε, αναθεώρηση της ναύτα, μήπως αυτές οι διαπραγματεύσεις έχουν, ε, επηρεάζουν και τις δικές μας διαπραγματεύσεις. Και τέλος, όσον αφορά τις επενδύσεις, το, το σύστημα το σύστημα το δικαστικό που θα δημιουργηθεί και την, για την προστασία των επενδύσεων. Μπορείτε να μας ενημερώσετε σε σχέση με αυτό το θέμα λίγο περισσότερο. Ευχαριστώ πολύ για την ΓΚΟΕ η κυρία Λόλα Σάντσες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όλοι συμφωνούμε με την μεγάλη ανησυχία που εκφράστηκε για την δραματική κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μεξικό, που διέρχεται ε, μία από τις πιο αιματηρές ε, περιόδους της ιστορίας του. Το 2000 ε, σκοτώθηκαν 70 άτομα τη μέρα. Είναι μία από τις χειρότερες χρονιές. Μιλάμε για δολοφονίες ακτιβιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοσιογράφων. Είναι ανησυχητική η κατάσταση αυτή και η ατιμορρησία στη χώρα. Επίσης, ε, ε, η, Μα, η Μαουρίτσια Πατρίθιο, ε, που είναι η πρόεδρος των Ιθαγενών του Μεξικού, δέχτηκε επίθεση όταν ταξίδευε σε ένα λεωφορείο στη χώρα. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε επιγόντως αυτό το πρόβλημα. Έχουν γίνει ουσιαστικές πρόοδοι τα τελευταία χρόνια. Και βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτω ώστε να μπουν αυτά τα κεφάλαια στι εμπορικέ συμφωνίε. Όπω είπαμε και την περασμένη εβδομάδα στην Ολομέλεια του Στρασβούργου, ε, θα πρέπει όμω να είμαστε πιο φιλόδοξοι και να εγγυηθούμε ότι είναι υποχρεωτικό να τηρούνται οι ρήτρε ε, των κεφαλαίων αυτών που αφορούν αυτά τα θέματα. Επίση, οι μηχανισμοί κυρώσεων είναι το μοναδικό εργαλείο που μπορεί να μας εξασφαλίσει ότι η προστασία αυτών των ρητρών θα είναι πραγματικά αποτελεσματική. Είναι σημαντικό επίσης να υπάρχει και μια ρήτρα αναθεώρησης του συνόλου της συμφωνίας. Η επικαιροποίηση του, της συμφωνίας αν δεν έχει αυτά τα στοιχεία που θεωρούμε ότι είναι ο ελάχιστος κοινός πανομαστής για να εξορροπήσουμε τις επιπτώσεις ε, της συμφωνίας και τις ασύμετρες επιπτώσεις που θα έχει, δεν θα μπορέσουμε σε καμία περίπτωση να την ε, υποστηρίξουμε. Ε, μία από τις βασικές κυρώσεις ε, Μάλλον θα υπάρχουν συγκεκριμένες κυρώσεις στην ε, συμφωνία και η ρήτρα αναθεώρηση θα υπάρχει επίσης. Για το περιεχόμενο των κεφαλαίων θα ήθελα να μου πείτε ε, ποια στοιχεία από τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα θα μπουν εκεί πέρα και επίσης ε, διάφορα στοιχεία ε, και διάφορες ρήτρες του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας δεν έχουν επικαιροποιηθεί και δεν έχουν γίνει, δεν τις έχει προσυπογράψει το Μεξικό. Θα μπουν στη συμφωνία αυτή. Επίσης, μην ξεχνάτε ότι όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνει η συμφωνία είναι πάρα πολύ ευραία και είναι πολύ σημαντικά για τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό θα πρέπει οι κυβερνήσεις των κρατών μελών θα, να, θα πρέπει να μπορούν να πούν τη γνώμη τους για αυτή τη συμφωνία. Γι' αυτό ε, οι, συμφω... ερωτήσεις μου είναι, ε, η συμφωνία αυτή θα μας δίνει αυτή τη δυνατότητα, θα είναι μια τέτοια μεικτή συμφωνία ε, όπως ονομάζεται. Η κυρία Χάουτολ από τους Πράσινους. Ευχαριστώ. Θέλω να θέσω δύο θέματα. Μιλήσαμε λίγο για την υποτελέμηση της διαφοράς και το, και το αντίστοιχο κεφάλαιο. Εγώ παραμένω επιφυλακτική. Γιατί μου φαίνεται ότι αυτό που προτείνεται δεν υπερβαίνει το επίπεδο των ε, εθελοντικών συστάσεων. Εγώ θα ήθελα να υπάρχει μια δυνατότητα επιβολής των μέτρων πολέμης διαφοράς εντός της συμφωνίας. Και δεύτερο θέμα. Ε, θα ήθελα να μάθω πώς προχωρούν οι διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της ναύτα και αν υπάρχει ενδεχομένως κάποια θεμελιώδης ε, διαφορά όσον αφορά την προσέγγιση που ακολουθείτε. Αφενός ε, στην ναύτα, είπα Καναδάς, Μεξικό αφενός και από την άλλη πλευρά, αφετέρου δηλαδή, στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Μεξικού και Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί αυτό μπορεί να είναι αποκαλυπτικό και ως προς τις μελλοντικέ διαπραγματεύσεις που θα έχουμε εμείς με τις ΗΠΑ. Ευχαριστώ. Ε, η κυρία Φάνερχάτς. Ευχαριστώ θεωρώ και εγώ ότι είναι πολύ σημαντικό να επικαιροποιηθεί μετά από 15 χρόνια η εν λόγω συμφωνία, αλλά συμφωνώ και εγώ ότι η ποιότητα έχει προβάδισμα έναντι της ταχύτητας. Γι' αυτό και θέλω να ρωτήσω. Τι θα γίνει με την εντολή διαπραγμάτευσης, θα δημοσιευθεί, θα μας γνωστοποιηθεί, γιατί θέλουμε και εμείς ως ευρωβουλευτές να γνωρίζουμε ακριβώς ποιο είναι το περιεχόμενο της εντολής για να μπορούμε και να, τηρήσουμε, και να διαμορφώσουμε τη στάση μας. Δεύτερον, για το σύστημα ICS που μας είπατε κι εσείς ότι υπήρχαν πολύ μεγάλες συζητήσει και προβλήματα. Ας μην το κρύβουμε. Ποια είναι η στάση του, του Μεξικό και ποια είναι η πρόοδος που έχει σημειωθεί. Διαφθορά. Μου φαίνεται ότι το συζητούμε αυτό το θέμα. Το ερώτημά μου όμως είναι αν δεν ε, τηρήσει τα συμφωνηθέντα το Μεξικό, ποια μέτρα θα λαμβάνονται. Και τελευταίο ερώτημα. Επειδή ε, ε μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το ζήτημα της βιωσιμότητας. Ε, είναι πολύ σημαντική οι μηχανισμοί κυρώσεων που θα προβλέπονται σε αυτή την συμφωνία. Γι' αυτό και πρέπει να συζητηθούν, καταρχά να θεσπιστούν στη συμφωνία και να προβλέπονται. Και θέλω να σας ρωτήσω συγκεκριμένα για αυτό το ζήτημα ποιε είναι οι συζητήσει που έχετε κάνει για αυτό το θέμα. Κύριε Μινουέρ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η Κομισιόν συνάπτει διάφορες συμφωνίες ελευθερών συναλλαγών σε όλο τον κόσμο και οι συγκεκριμένε διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν, επαναξεκίνησαν μόλις τον Νοέμβριο. Αλλά σε άλλες περιπτώσεις διαπραγματεύσεων της Ευρωπαϊκή Ένωσης ε, έχουμε διαπιστώσει οι μελέτε επιπτώσεων να διεξάγονται εκ των υστέρων, αφού δηλαδή έχουν υπογραφεί οι συμφωνίες. Επομένως, η μελέτη επιπτώσεων που αφορά τη συγκεκριμένη συμφωνία ε, δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει και διαβουλεύσεις ε, με ακτιβιστές ή οργανώσεις προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή του περιβάλλοντος. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Το Μεξικό έχει βεβαίω ε, κακή φήμη όσον αφορά την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναφέρθηκαν και ορισμένα από του συναδέλφου. Υπάρχουν ε, και συγκεκριμένε διεθνεί αναφορέ ω προ τη μεταχείριση που επιφυλάσσει το Μεξικό σε πρόσφυγε, ε, που είναι πάρα πολύ ανησυχητικέ. Όλα αυτά τα θέματα δεν είναι ε, θέματα που θα πρέπει να συμπεριληφθούν στι διαπραγματεύσει. Τι συμβαίνει λοιπόν με το συγκεκριμένο εγχειρίδιο που έχει εκδώσει η ίδια η Κομισιόν όσον αφορά τον, τη διαδικασία σύναψης και υπογραφής συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών. Αν πραγματικά πιστεύετε κι εσείς σε αυτό το εγχειρίδιο που εσείς οι ίδιοι έχετε συντάξει, μήπως θα έπρεπε να το χειρίζεστε με μεγαλύτερη σοβαρότητα. Ευχαριστώ πολύ. Και μένα... Δυο, δυο τρία επιπλέον σημεία. Η Έμα Κλάρκιν έθεσε το θέμα της ναύτα. Θα μπορούσατε να μας εξηγήσετε λιγάκι τις εξελίξεις, οι διαπραγματεύσεις που γίνονται στα πλαίσια της ναύτα, πώς επηρεάζουν τις δικές μας σχέσεις με το Μεξικό και κυρίως τα τελευταία νέα για τις διαπραγματεύσεις της ναύτα που ακούσαμε. Μπορεί να επηρεάσουν καθόλου τη στρατηγική της μεξικανικής πλευράς. Δεύτερον, το κεφάλαιο TSDT. Ξέρετε ότι στο Κοινοβούλιο έχουμε κάνει τεράστιες συζητήσεις για αυτό το θέμα. Μπορείτε να κάνετε μια επισκόπηση για το κεφάλαιο αυτό και αν το συγκρίνετε με το αντίστοιχο κεφάλαιο συμφωνία ΣΕΤΑ. Υπάρχουν εκεί κάποια καλά στοιχεία. Ότι οι εταίροι θα πρέπει να εγγυώνται ότι το εθνικό δικαστικό σύστημα είναι έτοιμο ούτω ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να διεκδικούν τα δικαιώματά τους εάν υπάρχουν παραβιάσεις στα πλαίσια του κεφαλαίου ε, TSDT ε, και να προσφεύγουν στα δικαστήρια. Για να συγκρίνουμε λοιπόν τα δύο αυτά κεφάλαια στην ε, Συμφωνία του Μεξικού ε, από τη μία ε, και στη συμφωνία, με το Μεξικό μάλλον και στη συμφωνία με, με τον Καναδά, στη ΣΕΤΑ. Κυρία Κιόνικ, ευχαριστώ. Πολλές ερωτήσεις μου υποβάλατε. Να ξεκινήσω με ένα σχόλιο που έγινε στην αρχή. Ε, για την ε, φιλοδοξία που θα πρέπει να διέπει αυτή την ε, συμφωνία. Φυσικά, ο στόχος μας είναι να έχουμε το ίδιο επίπεδο με την συμφωνία που προσυπογράψαμε πρόσφατα, τη ΣΕΤΑ. Και μην ξεχνάτε ότι και έχουν, ξεκινήσει παράλληλα και διαπραγματεύσεις στα πλαίσια τη ΝΑΦΤΑ, Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδάς. υπάρχουν και αντίστοιχε συμφωνίε όπως με, το, με Βιετνάμ και την Ιαπωνία. Τώρα, για τις δημόσιες προμήθειες. Είπα στην αρχή ότι η πρόσβαση σε, στην υπομοσπονδιακή αγορά είναι βασικό θέμα για μας. Το συζητάμε μακρόν με τους Μεξικανούς. Οι Μεξικανοί ποτέ δεν άνοιξαν την αγορά τους σε υποομοσπονδιακό επίπεδο για τις ε, δημόσιες προμήθειες αυτό το επίπεδο. Η κυβέρνηση θα πρέπει να κάνει ε, διαβουλεύσεις με τη συγκεκριμένη πολιτεία στο Μεξικό για να γίνει κάτι τέτοιο. Έχουν γίνει πάρα πολλές συζητήσει και σε υπουργικό επίπεδο και το θέμα αυτό και μπορούμε να πούμε ότι το Μεξικό έχει δεχθεί την αρχή τουλάχιστον του να συμπεριληφθούν και αυτά τα επίπεδα, τα υπόμοσπονδιακά δηλαδή, σε πολιτιακό επίπεδο στις στο κεφάλαιο των προμηθειών. Τώρα, με ποιο τρόπο είναι πιο επικίνδυνο, γιατί θα πρέπει να γίνουν ε, διαβουλεύσεις μεταξύ κράτους και πολιτείας. Είναι από τα κεφάλαια το, ε, από τα οποία δεν έχουν κλείσει ακόμα. Ε, είμαστε σε συζητήσεις υψηλού επίπεδου γι' αυτό και φυσικά το Μεξικό προσβλέπει και επιθυμεί να βρει κάποιους τρόπους για να γίνει δυνατό αυτό πριν ολοκληρωθεί ε, η συμφωνία. Τώρα για το διεθνές σύστημα, το διεθνές δικαστικό σύστημα, ε, το Δεκέμβριο συναντήθηκε η Επίτροπος Μάστροπ με τον, ε, με τον Υπουργό Γκουαχάλντο, ο οποίος είχε πει ότι το Μεξικό έχει δεχτεί να συνεργαστεί με το και να δεχτεί το νέο μας μοντέλο για τα επενδυτικά δικαστήρια που είναι ένα μεγάλο βήμα, ε, μια πρόοδο σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο ISTS ε, το οποίο ακολουθούσε ε, το Μεξικό σε όλες τις διμερείς συμφωνίες του. Επίσης, συζητάμε και το πολυμερές επενδυτικό δικαστήριο. Φυσικά δεν είναι ο στόχος εδώ να συμπεριληφθεί αυτό το πολυμερές επενδυτικό δικαστήριο στην συμφωνία είναι κάτι που εκφεύγει τις συμφωνίες, αλλά υπήρχε ενδιαφέρον από το Μεξικό και για αυτό το θέμα, γιατί υπάρχουν και οικονομικές επιπτώσεις. Αν μπορέσεις, δηλαδή, να περάσεις από ένα διμερές σύστημα σε ένα πολυμερές σύστημα, φυσικά θα έχει οικονομικές επιπτώσεις. Όμως, για αυτή τη φάση των διαπραγματεύσεων επικεντρωνόμαστε στο διμερές επενδυτικό δικαστήριο και στις σχετικές διατάξεις, ε, και είμαστε ακόμα σε φάση συζήτησης γι' αυτό, για τις γεωγραφικές ενδείξεις. Ναι. Υπάρχουν κάποια καθόδη θέματα. Συνδέεται με την πρόσβαση στην αγορά για τα γεωργικά προϊόντα. Το Μεξικό πρέπει να ξέρετε ότι ετοιμάζει μια εσωτερική νομοθεσία για τις ε, γεωγραφικές ενδείξεις εδώ και χρόνια. Από τις τελευταίες εμπορικές συμφωνίες μας θα ξέρετε επίσης ότι η δική μας πλευρά επιμένει πολύ όλοι ότι όλες οι βασικές γεωγραφικές ενδείξεις από το δικό μας κατάλογο να προστατεύονται στο Μεξικό θα θυμάστε επίσης ότι κανονικά υπάρχουν καμιά δεκαριά γεωγραφικές ενδείξεις ε, που είναι υποσυζήτηση όπου προσπαθούμε να έχουμε διαφορετικά επίπεδα ευελιξίας. Το κάναμε αυτό και στη ΣΕΤΑ, το κάναμε και με την Ιαπωνία. Και αυτό σας δείχνει ότι εκεί όπου υπάρχουν τα πραγματικά οικονομικά και εμπορικά συμφέροντά μας, η δική μας πλευρά προσπαθεί να βρει λύσεις, είναι έτοιμη να βρει λύσεις. Φυσικά θα πρέπει να έχουμε καλά επιχειρήματα ε, σε, που να εδράζονται σε, οικονομικά, σε οικονομική βάση και νομική βάση ούτως ώστε να μην έχουμε γραφικές ενδείξεις που είναι απροστάτευτες για την ε, εντολή. Όπως θα ξέρετε κατά πάσα πιθανότητα, η Κομισιόν θα πρέπει να ζητήσει την εντολή για το Μεξικό και τις διαπραγματεύσεις ε, και να ζητήσει να δημοσιευθούν αυτά τα θέματα, η διεντολή δηλαδή. Δεν έχω νέα για αυτό το θέμα. Ε, έχει δημοσιευθεί πρόσφατα η σχετική εντολή για την συμφωνία με τη Χιλή. Θα ζητήσουμε να... Έχουμε ζητήσει να δημοσιευτεί και η εντολή για το Μεξικό. Για τα βασικά εναπομείναντα θέματα, για τις ζωφικές ενδείξεις ε, μόλις αναφέρθηκα και σε προηγούμενες παρουσιάσεις μου έχω πει ότι υπάρχουν διάφορα θέματα πρόσβαση στην αγορά γεωργικών προϊόντων όπου πρέπει να συζητήσουμε και να συμφωνήσουμε το επίπεδο των ε, δασμών. Και αυτές οι διαπραγματεύσεις προφανώς είναι αλληλένδετες, όλα τελικά είναι ένα πακέτο, γιατί δεν πρόκειται να συμφωνήσουμε τίποτα αν τα συμφωνήσουμε όλα. Όλα είναι επιτάπητο. Θα γίνουν ε, λοιπόν περισσότερες συζητήσεις επόμενε εβδομάδες και νομίζω ότι το Μεξικό ξεκαθάρισε ότι ενδιαφέρεται πάρα πολύ για θέματα πρόσβασης στην αγορά και εμείς προφανώς, αλλά εμάς μα ενδιαφέρουν και γραφικές ενδείξει. και κάποια από τα βασικά κεφάλαια για τους κανόνες ICS, δηλαδή το Διεθνές Δικαστήριο κτλ, ε, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας κτλ. Για το TSD. Αυτό ε, το κεφάλαιο τώρα στην συμφωνία με το Μεξικό είναι ανάλογο με τη συμφωνία ΣΕΤΑ τσεκάρουμε τι συμφωνήσαμε στους τελευταίους γύρους, το τελευταίο γύρο το Δεκέμβριο. Αυτό το ε, κείμενο θα έρθει ενώπιον του Κοινοβουλίου σύντομα. Στη σύμβαση του ILO, του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, το βασικό είναι να εφαρμόζεται η σύμβαση, ε, την οποία έχουν, ε, σε περίπτωση που την έχουν προσυπογράψει και δύο πλευρές και την έχει προσυπογράψει το Μεξικό και θα προσπαθούμε κάθε φορά να επικυρώνονται οι συμφωνίες του ILO που δεν, όταν δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Για την εφαρμογή του κεφαλαίου TSD ε, είναι... το συζητάμε εδώ στο Κοινοβούλιο το θέμα αυτό, αλλά δεν το συζητάμε στις διαπραγματεύσεις. Για την συμφωνία με το Μεξικό προβλέπεται μία ρήτρα αναθεώρησης αντίστοιχη με αυτή που έχουμε και στη ΣΕΤΑ γιατί οι συζητήσεις εσωτερικά δεν έχουν οριστικοποιηθεί για αυτό το πολύ επίκαιρο θέμα και για το θέμα των ε, κυρώσεων. Και προς το παρόν είναι πρόωρο πριν οριστικοποιηθούν αυτές οι συζητήσεις να μπει στο κείμενο υπο, που είναι υποδιαπραγμάτευση. Τώρα, ένα άλλο κεφάλαιο για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Ένα κεφάλαιο ανοιχτό, συζητάμε το μηχανισμό, συζητάμε το πώς θα το επιβάλλουμε. Ε, δεν μπορώ να το σχολιάσω σε αυτή τη φάση. Φυσικά η Κομισιόν θέλει την πιο ισχυρή δυνατή δέσμευση, αλλά δεν μπορώ να δεσμευτώ για το που θα καταλήξουμε στο κεφάλαιο αυτό για τη διαφθορά. για το ζήτημα των δύο φύλων. Το θέμα αυτό δυστυχώς αναδείχθηκε κάπως αργά στην πορεία των συζητήσεων. Δεν το έχουμε λοιπόν παρουσιάσει επισήμως ακόμα στο Μεξικό. Δεν ε, εντασσόταν στα θέματα που είχαμε σκοπό να συζητήσουμε. Βεβαίως ε, το ζήτημα αυτό καλύπτεται υπό την πολιτική συμφωνία. Γι' αυτό και θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε όταν θα περάσουμε, τι, μπορούμε να κάνουμε στη φάση της ε, εφαρμογής αυτής της συμφωνίας σε συνεργασία με το Μεξικό γιατί βεβαίως υπάρχει ε, η Γενική Συμφωνία, η Παγκόσμια Συμφωνία και αυτή η συμφωνία θα αποτελέσει βεβαίως τμήμα αυτής. Εκεί λοιπόν βεβαίως υπάρχουν ζητήματα που μπορούν να συζητηθούν υπό τον μηχανισμό πολιτικής ε, εφαρμογής. Όσον αφορά τη Συμφωνία των Παρισίων, πρόκειται για ένα θέμα στο οποίο επιμένουν διάφορες πλευρές, ε, ιδίως η Γαλλία, όμως και αυτές οι συζητήσεις ε, έφτασαν λίγο αργά και δεν θέλουμε τώρα να εμποδίσουμε την ε, υπογραφή, την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία αυτή. Μόλις όμως κλείσει το κεφάλαιο, είναι, καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολο να ξαναξεκινήσεις από την αρχή τη συζήτηση για να προσθέσεις ένα καινούριο θέμα. Κάτι τέτοιο θα πάρει την, ε, την ε, διαδικασία. Για το SIA θα θυμάστε ότι η Κομισιόν διεξήγαγε μελέτη επιπτώσεων πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Η συγκεκριμένη διαδικασία αξιολόγησης βιωσιμότητας προηγήθηκε της έναρξης των διαπραγματεύσεων. Είναι δύσκολη διαδικασία. Ε, είναι χρονοβόρα διαδικασία και δαπανηρή. Και ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε, μια από τις προκλήσεις που είχαμε σε σχέση με αυτές τι διαπραγματεύσει ήταν ότι θέλαμε να ολοκληρωθούν γρήγορα, σε περίπου 1,5 χρόνο. Και παρά το γεγονός ότι καταβάλαμε όποια προσπάθεια ε, μπορούσαμε, δεν ήταν δυνατόν ποτέ μια τέτοια μελέτη επιπτώσεων όσον αφορά τη βιωσιμότητα να ολοκληρωθεί μέσα σε ένα τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Βεβαίω, έχουμε υπόψη μα και τι διάφορε εκθέσει που έχουν δημοσιευθεί παρά το γεγονός ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η τελική έκθεση, δεν έχει δημοσιευθεί ε, και έχουμε συζητήσει το θέμα αυτό και στο πλαίσιο της κοινωνίας των πολιτών θα γίνει και μια ακόμη συζήτηση εντός του Φεβρουαρίου για την επόμενη έκθεση που θα συνταχθεί που επίσης δεν θα είναι η τελική αλλά ελπίζουμε την τελική να την ετοιμάσουμε πριν από το καλοκαίρι. Πιστέψτε με, εγώ προσωπικά λυπάμαι που δεν έχουμε καταφέρει να την ολοκληρώσουμε αυτή την μελέτη. Δυστυχώς όμως είμαι ειλικρινής. Δεν ήταν εφικτό να ε, περάσουμε από όλε τι διαδικασίες που προβλέπονται για το SIA και να, και να δημοσιεύσουμε και μια οριστική έκθεση. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν λαμβάνουμε υπόψη μας όλα αυτά τα στοιχεία στις διαπραγματεύσεις μας. Ευχαριστώ. Ίνμα, θέλεις να κάνεις τις καταληκτικές παρατηρήσεις. Ναι, πολύ σύντομα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη της ΣΥΝΤΑ για την συμμετοχή και το ενδιαφέρον είμαι βεβαία ότι θα δουλέψουμε αρμονικά. Ήταν πολύ χρήσιμο που η Κομισιόν μπόρεσε να έρθει και να μας ακούσει. Είναι σημαντικό λοιπόν να προχωράμε σε αυτές τις νέες εμπορικές συμφωνίες που περιλαμβάνουν ε, ρήτρε στο κεφάλαιο της βιώσιμης ανάπτυξης, οι οποίες να είναι αποτελεσματικές, να είναι εφικτές και να μπορεί να εσωματώνεται και ένας μηχανισμός ε, κυρώσεων Δεν έχουμε διευκρινίσει ακριβώς ποιος θα είναι ο μηχανισμός με όλες τις λεπτομέρειες, αλλά θα πρέπει να ξέρουμε πώς θα το εφαρμόσουμε. Είναι πολύ σημαντικό. Αυτές οι πτυχές μας ανησυχούν περισσότερα, ε, όπως η διαφθορά που είναι το βασικό στοιχείο που πρέπει να καταπολεμήσουμε, γιατί διαφορετικά είναι πολύ δύσκολο να ξέρουμε πώς θα μπορούμε να βοηθήσουμε με μια εμπορική συμφωνία ώστε να ε, καταπολεμήσουμε αυτήν την μάστιγα και έπειτα για την ε, Συμφωνία Πολυμερών ε, Επενδύσεων. με το Καναδά είχαμε ακολουθήσει αυτή τη συμφωνία, είχαμε ακολουθήσει αυτό το πρότιμο. Θα πρέπει οι χώρες να μπορούν ε, να χρησιμοποιούν ένα μοντέλο το οποίο να συμβάλλει στην επίλυση του προβλήματος της λύσης διαφορών σε πολυμερές επίπεδο, σε επίπεδο κρατών επενδυτών. Νομίζω πως εδώ είναι πολύ σημαντικό και θα πρέπει οι διαπραγματευτές να λάβουν λάβουν υπόψη τι λέει αυτό εδώ το κοινοβούλιο, γιατί αυτό το κοινοβούλιο εδώ θα πρέπει να ψηφίσει τελικά και να εγκρίνει και αντιπροσωπεύουμε την υπεράσπιση των συμφερόντων όλων των ε, πολιτών. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ και έτσι ολοκληρώνεται το σημείο 13 και στρεφόμαστε στο σημείο 14 της ημερησίας μας διάταξης. Πρόκειται για τη συνεχιζόμενη διαπραγμάτευση που προχωράει όμως λίγο πιο αργά γιατί ο εταίρος είναι η Ινδία. Ξεκινήσαμε τις διαπραγματεύσεις το 2007. Είναι μια συνεχής διαδικασία. Ένα από τους κεντρικούς μας διαπραγματευτές, ο κύριος Κένιγκ, είναι εδώ μαζί μας και ε, συμμετέχει και στις διαπραγματεύσεις με την Ινδία και ο πρέσβης της Ινδίας, ο κ. Κούμα, ε, καλωσορίσατε. Είναι παρόν να αρχίσουμε λοιπόν με την κυρία Κούνιγκα και μετά να δώσω το λόγο στον κύριο Κούμα. Ο εισηγητής μας είναι ο κύριος ε, David Κάμπερ. Κυρία Κένιγκ, σας ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Μεγάλη μου χαρά που είμαι σήμερα εδώ και βεβαίως ε, την παρουσία της ε, εξοχότητας κυρίας Κούμα και μιλώ εξ ονόματος της Επιτροπής, Επιτροπής. Είναι καλή ε, χρονική στιγμή για να ε, κάνουμε μια ε, ε, να σας δώσουμε μια εικόνα για τις διαπραγματεύσει και το πού βρισκόμαστε. Όπως τόνισε ο Πρόεδρος, ε, έχω, δεν είχαμε επίσημος γύρους διαπραγματεύσεων από το 2013. Ωστόσο, έχουν γίνει αρκετές συζητήσεις για τις προοπτικές, για την έναρξη, επανέναρξη μάλλον των διαπραγματεύσεων και αυτό νομίζω πως είναι πολύ επίκαιρο γιατί μόλις τελείωσε η διάσκεψη κορυφής του Οκτωβρίου στο Δελχή του περασμένου έτους και σε αυτή τη διάσκεψη κορυφής η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, προηγήθηκε και ο Πρωθυπουργός ε, της χώρας ε, διαπίστωσε τις προσπάθειες επανέναρξης. Μεγάλη δέσμευση δόθηκε στη σημασία ενίσχυσης των εμπορικών σχέσεων ανάμεσα στην Ένωση και την Ινδία και θα ήθελα να ξεκινήσω με αυτό ότι δηλαδή δεν υπάρχει καμιά δισταγμός όσον αφορά ακριβώς αυτό την ενίσχυση των εμπορικών σχέσεων. Συζητήσεις για την ε, Συμφωνία Ελευθέρου Μπορείου είναι το ένα μέρος αυτού, ένα σημαντικό μέρος αυτού, μόνο που έχουμε δει από το 2013 ε, συνεχίσει τις διμερείς μας συζητήσεις για διάφορα ζητήματα. Έχουμε τακτικές ε, συνεδριάσεις των ομάδων εργασίων μας που έχουν φέρει καρπούς, δηλαδή δεν είναι όλα σε λανθάνουσα κατάσταση. Ε, μετά από την ε, διάσκεψη κορυφής του Οκτωβρίου αποφασίστηκε ότι οι δύο κύριοι διαπραγματευτές, εγώ δηλαδή και η κυρία Άννητα Παβένα θα είχαμε επαφές και όντως είχαμε επαφές τον Νοέμβριο στο Δελχή όπου διατρέξαμε διάφορα κεφάλαια όπου είχαμε σημαντικές πολιτικές εξελίξεις στη διάσταση όπως αυτή που ανέφερα και για το Μεξικό πριν από λίγο ότι έγιναν πολλές αλλαγές τα τελευταία χρόνια από την άποψη της Ένωσης ισχύει αυτό όταν μιλάμε για διαπραγματεύσεις έχουν υπάρξει και διάφορες αλλαγές που πρέπει να αντικατοπτρίζονται σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση όταν, όταν δηλαδή θα αρχίσουμε να εξετάζουμε, να σκεφτόμαστε πόσος χρόνος έχει περάσει. SPS, TBT, δημόσιες προμήθειες, IOP, πνευματικά και η εμπόριο και βιώσιμη ανάπτυξη, Έχουμε όλο και περισσότερη σαφήνεια για τις διαφορές που έχουμε και για το τι μπορεί να είναι εφικτό μέσα στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων. Αυτό λοιπόν που αποφασίσαμε μετά από αυτή τη συζήτηση ήταν ε, ότι θα έπρεπε σε τεχνικό επίπεδο να συνεχίσουμε να διερευνούμε ε, πού μπορούσε να υπάρξει ε, διαφορά. Είναι σημαντικά θέματα, θέματα κλειδιά, κεφάλαια κλειδιά και η επικεφαλής των διαπραγματεύσεων τα θέλαν να ε, μιλήσουν και πάλι ε, για να δούμε ακριβώς πού βρισκόμαστε, να κάνουμε μια αξιολόγηση, να πούμε ποιες είναι οι συστάσεις μας, να συνοψίσουμε και πάλι τις διαπραγματεύσεις, εάν όντως υπάρχει μια τέτοια δυνατότητα, αλλά να μπορέσουμε να δώσουμε και στα κράτη-μέλη και σε άλλους φορείς να γνωρίζουν τι μπορούν να περιμένουν, εάν επαναληφθούν οι διαπραγματεύσεις. Ένα ιδιαίτερο θέμα βεβαίως, το οποίο συζητείται εδώ και αρκετά χρόνια, είναι η προστασία των επενδύσεων και αυτό το κομμάτι της συμφωνίας. Και εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι είναι κομμάτι των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων και η Ινδία επιμένει πολύ ώστε αυτό να μείνει μέσα στις διαπραγματεύσεις. Θα θυμάστε ίσως αξιότιμοι κύριοι Ευρωβουλευτές ότι στα τέλη του 2005 συμφωνήσαμε για ένα νέο μοντέλο για την προστασία των επενδύσεων και το στείλαμε στην, στα κράτη-μέλη. Βεβαίω, τότε η Κομισιόν τόνιζε πω θα ήταν πιο ωφέλιμο να διατηρηθούν αυτέ οι προστασίε μέχρι ότου να έχουμε μια, ένα νέο σύστημα επενδυτικού δικαστηρίου. Αλλά δυστυχώς έκτοτε έχουν εκπνεύσει οι περισσότερες διμερείς ε, συμφωνίες. Υπάρχουν κάποιες ε, ομοιότητες ανάμεσα στις προηγούμενες διμερείς ε, συμφωνίες για την επίλυση των διαφορών και την ε, προτινόμενη λύση του επενδυτικού δικαστηρίου, δυνατότητα δηλαδή Ε, να περανάν αυτές οι διαφορές στο πολυμερές επίπεδο. Υπάρχουν όμως κάποιες διαφορές όπως ας πούμε η εξαίρεση των φόρων, το αίτημα για την εξαίρεση των φυσικών ε, φαρμάκων ε, και διάφορα άλλα, και διάφορες άλλες λεπτομέρειες. Το συζητάμε και από τις δύο πλευρές για να προσπαθήσουμε να δούμε πού είναι πιο ευέλικτος ο καθένας, αλλά υπάρχουν και πολλές προκλήσεις. Όπως είπα, έχουμε και έναν απολογισμό που προβλέπουμε να κάνουμε στις αρχές του Απριλίου και να δούμε ε, κάποιες ε, κατευθυντήριες γραμμές για την επόμενη διάσκεψη κορυφής που δεν έχει ακόμα καθοριστεί η ημερομηνία, αλλά αναμένουμε να γίνει εδώ στις Βρυξέλλες κάπου το φθινόπωρο. Ευχαριστώ πολύ. Πρέζης Κούμα, παρακαλώ. Σας, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλα τα μέλη ε, του Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να μοιραστώ μαζί σας τις πληροφορίες που έχω. Ευχαριστώ την επικεφαλή των διαπραγματεύσεων που έδωσε μια πολύ ξεκάθαρη εικόνα για το πού βρισκόμαστε Στη 14η διάσκεψη κορυφής οι κοινέ δηλώσεις που έγιναν κατέστησαν σαφές και έδωσαν σαφή μηνύματα και από, από τους ηγέτες μας ότι είναι προσιλωμένοι στην προσπάθεια επανέναρξης των διαπραγματεύσεων για μια ολοκληρωμένη και αμοιβαία ε, εποφελή εμπορική συμφωνία. Βεβαίως η Ινδία ήταν και είναι, παραμένει έτοιμη να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις, αλλά καταλαβαίνουμε ότι η ευρωπαϊκή πλευρά είχε συγκαλέσει, ε, μάλλον μας είχε ενημερώσει εκείνη τη συνεδρίαση και ότι θα έπρεπε να ισχύουν κάποιες προϋποθέσεις, δηλαδή οι προδιαπραγματεύσεις για τον τρόπο με τον οποίο ε, θα προχωρήσουμε γίνονται. Όπως ανέφερε και η επικεφαλής των διαπραγματεύσεων, ε, έγινε ένας καλός γύρος διαπραγματεύσεων τον Νοέμβριο και έχουν γίνει και επαφές ε, μεταξύ των διαφόρων αρμοδίων οι ηγέτες ε, που έχουν ε, θεσπίσει 13 άξονες πορείας μας έδωσαν τις κατευθυντήριες γραμμές. Επόμενη, ε, Επόμενη μάλλον επαφή ε, είναι προγραμματισμένη για τον Απρίλιο. Η Ινδία θα ήθελε να, γίνει, να, να, να ξεκινήσει έγκαιρα και να ολοκληρωθεί έγκαιρα μια συμφωνία όπου εξετάζονται οι εμπορικές αλλά και οι επενδυτικές σχέσεις. Εγώ ήμουν στο Δελχή αυτόν τον Ιανουάριο και μετά, τώρα, αφού, μετά από τις επαφές μου με τις αρχές, έχω κάθε λόγο να ελπίζω πως θα σημειωθεί σημαντική πρόοδος φέτος για την επανέναρξη, όπως ελπίζουμε, των ίδιων των διαπραγματεύσεων. Να διευκρινίσω ότι όταν οι δύο μετά από υπουργική αποφασία στείλανε ένα μήνυμα ότι θα θέλαμε να πάψουν οι ισχύουσες επενδυτικές συνθήκες με πάνω από 80 χώρες. Ε, αυτό συνέβη γιατί υπήρχαν κάποια προβλήματα στο κείμενο. Στείλαμε λοιπόν ένα πρότυπο κείμενο σε όλους, ε, επιμένουμε σε αυτό και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις από αυτού του κειμένου και με τα κρατημέλη. Αλλά βεβαίως το Ευρωπαϊκό Σύστημα λέει ότι θα πρέπει η ίδια η Ένωση να αρχίσει διαπραγματεύσεις, οπότε ήταν κάτι το γενικό, δεν είχε στόχο μόνο τα κράτη-μέλη. Ήθελα απλά να διευκρινίσω πως η λήξη των προηγούμενων συμφωνίων δεν σημαίνει το τέλος της προστασίας των επενδύσεων, γιατί υπάρχει μια ρήτρα sunset που προβλέπει την παράταση της προστασίας για όλες τις επενδύσεις για επιπλέον 15 με 20 χρόνια, ανάλογα με το η ρήτρα ε, ολοκλήρωσης των συγκεκριμένων συμφωνιών. Αυτή είναι μια διευκρίνηση λοιπόν. Είμαστε έτοιμοι, όπως σας είπα, να διαπραγματευτούμε συμφωνίες διμερείς για την προστασία των επενδύσεων, αν αυτό χρειαστεί, αλλά Σύμφωνα με τη συνθήκη της Λισαβόνας και τους κανόνες <coughs> της Ένωσης, η διαπραγματευτική αρμοδιότητα ε, ε, βαραίνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει ε, να κατανοήσετε ότι η, Ινδία είναι αναπτυσσόμενη χώρα με πολλούς τομείς προηγμένους, ενώ υπάρχουν και τομείς που έχουν μείνει πίσω, που, έχουν, που υστερούν μπορούμε σε πολλούς τομείς να είμαστε ελεύθεροι, ενώ είναι προς το, θυμόσιο, ε, το εθνικό μας συμφέρον όσον αφορά τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στο μεταπητικό τομέα. Πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί και γνωρίζουμε πώς από την πλευρά σας αναγνωρίζετε αυτές τις ιδιαιτερότητες. Ο Πρωθυπουργό μα, κύριε Πρόεδρε, είναι αποφασισμένο ότι θα πρέπει να συνεργαστούμε με την Ένωση για να φτάσουμε σε μια εμπορική και επενδυτική συμφωνία με τρόπο ώστε και οι δύο πλευρέ να βγουν κερδισμένες. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια και η Ινδία έχει επιφέρει αλλαγές στις πολιτικές της που βαραίνουν την στάση μας και την προσέγγισή μας προς τις διαπραγματεύσεις και πάνω απ' όλα είμαστε αποφασισμένοι να τα θέσουμε όλα αυτά σε εφαρμογή και να ε, το πετύχουμε. Οι επενδύσεις έχουν αυξηθεί, η Ένωση έχει δείξει ενδιαφέρον στο να συμμετέχει στις βασικές πρωτοβουλίες της Ινδίας, όπως η ψηφιακή Ινδία, ε, και αυτό το καλωσορίζουμε και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει φτιάξει γραφείο στο Νέο Δελχή. Είμαστε ευτυχείς γι' αυτό και ήδη έχουμε ξεκινήσει με τεράστια προγράμματα και πρωτοβουλίες. Επίσης θεσπίσαμε μια, έναν μηχανισμό ε, διευκόλυνσης των επενδύσεων στην ε, Ινδία ε, όπου μοιραζόμαστε τις καλύτερες πρακτικές και τις καινοτόμες τεχνολογίες. Το καλωσορίζουμε αυτό και σύντομα θα ανακοινώσουμε μια αναθεωρημένη βιομηχανική πολιτική. Έχουμε συντάξει και ένα νομοσχέδιο για την προστασία των ε, δεδομένων πιο ευθυγραμμισμένο με την ευρωπαϊκή πολιτική από ό,τι οποιοδήποτε άλλο άλλη πολιτική. Οπότε κύριε Πρόεδρε, ε, υπάρχει μια λογική που λέει ότι θα πρέπει λοιπόν να συνεργαστούμε ε, Ινδία με Ευρωπαϊκή Ένωση όσο γίνεται περισσότερο στους επόμενους μήνες και εγώ ως πρέσβης θα διευκολύνω τους διαπραγματευτές και από τις δύο πλευρές όσο περνάει από το χέρι μου. Ευχαριστώ πολύ. Ε, κύριε Ευχαριστώ Κυρία Πρέσβυρα, κυρία Κόνιχ, χαιρόμαστε που είστε μαζί μας. Εγώ μάλιστα έχω συστήσει στο παρελθόν και μια ομάδα παρακολούθησης. Δυστυχώς όμως δεν είχαμε και πολλά πράγματα να παρακολουθήσουμε. Φαίνεται ότι υπάρχουν κάποια θετικά σημεία προόδου, τα ακούσαμε και το πρωί, ιδίως σε επίπεδο τεχνικών εμπειρογνωμών. Και εδώ το χαιρετίζω αυτό. Όμως ε, νομίζω ότι είμαστε όλοι αρκετά απογοητευμένοι από την έλλειψη πρόοδου. Και όπως ακούσαμε ε, το τέλμα των διαπραγματεύσεων διαρκεί εδώ και πέντε χρόνια. Μιλάμε για μια αγορά 1,2 ε, δισεκατομμυρίων ανθρώπων με τεράστιες δυνατότητες, πολλές δεξιότητες, μεγάλη αγορά εργασίας. Έχουμε υψηλότερους δασμούς ε, στα είδη πολυτελείας, ε, ε, έχουμε εξαγωγές προς την Ινδία, αυτοκινήτων, σκοτζέζικου ουίσκι και όλα αυτά βεβαίως τα προβλήματα που υπάρχουν στις εμπορικές μας σχέσεις που δεν έχουν λυθεί ακόμα πλήττουν και τους Ινδούς αλλά και τους Ευρωπαίους και δεν, δεν εξαντλούνται τα, τα ζητήματα μόνο στη βιομηχανία. Μιλάμε και για τις δημόσιες προμήθειες, για τη φαρμακοβιομηχανία. Ε, νομίζω ότι χρειάζεται να υπάρξει μια πραγματική επανέναρξη των διαπραγματεύσεων που θα πρέπει να ξεκινήσουν ε, το συντομότερο δυνατό. Και εδώ τίθενται κάποια ζητήματα σε σχέση με το πώ θα προχωρήσουμε. Έχοντας υπόψη και το τι διεμήφθη στην υπουργική διάσκεψη στο Μπουένο Άιρε, νομίζω ότι εκεί εμφανίστηκε μια μη, μη επικοδομητική ε, προσέγγιση γενικά για το εμπόριο. Ίσως αυτό απαντά και στο γιατί έχει υπάρξει αυτή η καθυστέρηση. Η Ινδία πιστεύει στο ελεύθερο εμπόριο τελικά. Είναι κάτι που επιδιώκει και την ενδιαφέρει. Αυτό είναι ένα βασικό ερώτημα. Θα έλεγα λοιπόν ότι πρέπει να ξεκινήσουν σύντομα από την αρχή οι διαπραγματεύσει και χαίρομαι για τα όσα είπε η πρέσβυρα ως προς αυτό. Θέλω να πω και τα εξή. Προφανώς μιλούμε για Συμφωνία Επενδύσεων και Εμπορίου, BTIA. Έπειτα από την ε, απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τη Σιγκαπούρη πρέπει να σκεφτούμε θα μήπως θα ήταν καλύτερα να αφαιρεθούν να αφαιρεθεί η διάσταση των επενδύσεων από την συγκεκριμένη συμφωνία προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία ή θα συνεχίσουμε να διαπραγματευόμαστε και για, τις, και για τους δύο τομείς, και για τις επενδύσεις και για το ε, εμπόριο. Γιατί κάτι τέτοιο θα ερχόταν και σε αντίθεση με την απόφαση του δικαστηρίου. Άρα το ερώτημα είναι, θα αφαιρέσουμε τις επενδύσεις και δεύτερο ερώτημα. Πώ θα καταφέρουμε αυτή την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, Ποια είναι ακριβώ τα εμπόδια, Μήπω είναι θεμελιώδη ζητήματα προσέγγιση γενικά για το ελεύθερο εμπόριο, ή μήπω είναι απλούστερα τα θέματα που θα μπορούσαν και να λυθούν δηλαδή. Ε, να αρθούν αυτά τα εμπόδια που έχουν εμφανιστεί, αν είναι έτσι, προκειμένου να ξεκινήσει γρήγορα η διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι συμφωνούμε σε όλα αυτά, λέει ο Πρόεδρος. Πολλά μέλη της Επιτροπής ε, έχουν ζητήσει τον, ε, το λόγο και γι' αυτό ένα λεπτό καθένας και μόνο. Κάντε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την ενημέρωση αυτή. Θα ήθελα να χαιρετήσω την επικεφαλής ε, διαπραγματεύτριά μας, αλλά και την πρέσβερα την κυρία Κούμα. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά τα ζητήματα, ε, στο τι προγραμματίζεται, να υποβληθεί σε διαπραγμάτευση. Σε διαπραγμάτευση. Ε, νομίζω ότι ένα πρώτο βήμα θα ήταν να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια για την προστασία των επενδυτών. Θέλω να θέσω το εξή ερώτημα. Το νέο μοντέλο, το SWIT, ε, ποια είναι η άποψη της Κομισιόν για αυτό. Ε, εδώ έχει τεθεί το ζήτημα της, ε, της, της προστασίας των επενδυτών και προβλέπεται να εξαντλούνται πρώτα τα μέσα σε εθνικό επίπεδο προτού, μπορεί κανείς, προτού να μπορεί κανείς να προσφύγει σε ICTS για τη διαβιωσιμότητα. Η Ινδία γενικά δεν διαπραγματεύεται για κεφάλαιο βιωσιμότητα αυτή τη στιγμή. Θα συμφωνούσε όμω να προσθεθεί κάτι τέτοιο ακόμη και αν δεν περιλαμβάνονται πάρα πολύ αυστηρέ διατάξει και ρήτρε. Θα ήθελα πάρα πολύ να μάθω ποια είναι η θέση της Κομισιόν. Ε, θεωρεί ότι τα πρότυπα του ILO, για παράδειγμα, είναι ε, προϋποθέσεις για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων. Πώς το χειρίζεται το συγκεκριμένο ζήτημα. κυρία Ρόβολ. Ε, νομίζω ότι ε, πρέπει να... Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ε, κυρία Πρέσβηδα και την Κομισιόν για την πολύ ολοκληρωμένη ενημέρωση. Νομίζω ότι με κάποιον τρόπο χάσαμε την, τη δυναμική που είχε δημιουργηθεί πριν από κάποια χρόνια, γιατί σε τελική ανάλυση η Ινδία είναι η μεγαλύτερη δημοκρατία του κόσμου. Αυτό και μόνο ε, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας, όχι μόνο εμείς και οι Ινδοί, προκειμένου να ε, ξανατονώσουμε τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων. Θέλω να ε, ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο σχετικά με την προστασία των επενδύσεων είναι ένα θέμα που μας απασχολεί πάντοτε. Μετά την Λισαβόνα, βεβαίως ε, το θέμα αυτό αποτελεί αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταυτόχρονα όμως ισχύει ε, και οδηγία, η οποία εγκρίθηκε στην προηγούμενη νομοθετική θητεία, η οποία προβλέπει ότι ε, μπορούν να συνεχίσουν να ισχύουν και διμερείς συμφωνίες. Και πρέπει να πω, αν θέλουμε να δημιουργήσουμε μια δυναμική αυτή τη στιγμή, εγώ θα έλεγα ότι είναι αντιπαραγωγικό να καταργήσουμε συμφωνίες δημιουργίες, οι οποίες ε, σε κάποιο βαθμό, κάποιες από αυτές μάλιστα, ε, ισχύουν και αποφέρουν αποτελέσματα εδώ και πολλά χρόνια. Θα έλεγα λοιπόν ότι δεν πρέπει να είναι αυτό το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε. Η, ο εκπρόσωπος των, ε, της Γκουε έχει το λόγο. είστε. Κύριε Πρόεδρε, οι διαπραγματεύσει με την Ινδία ε, είχαν βρεθεί σε τέλμα για πολλά χρόνια. Ξεκίνησαν το 2007, αλλά φαίνεται ότι τελικά για πολλά χρόνια ε, υπήρξε, υπήρξε ένα πάγωμα των διαπραγματεύσεων. Ε, αλλά τα πράγματα αλλάζουν. Η Ινδία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και βεβαίως μια τέτοια συμφωνία με την ε, ε, Ινδία θα έχει και σημαντικές γεωπολιτικές επιπτώσεις. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω τα εξής. Η Κομισιόν τι ακριβώς έχει υποσχεθεί στην Ινδία προκειμένου να επανέλθουν στο τραπέζι των πραγματεύσεων. Υπάρχει ζήτημα με τις, ε, με τις υπηρεσίες. Ξέρουμε ότι στην Ινδία υπάρχει πρόβλημα ε, με τις υποχρεώσεις επισήμανσης αλλά και υγειονομικής προστασίας των, των τροφίμων συγκεκριμένα. Επίσης, ε, outsourcing στο διαδίκτυο. Πρόκειται για ένα κοινωνικό πρόβλημα. Είναι ένα ζήτημα που έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα σε εργαζόμενους σε ολόκληρο τον κόσμο. Γιατί στην Ινδία είναι γενικευμένο φαινόμενο να μην υπάρχει καμία προστασία των εργαζομένων. Τι θα κάνει η Κομισιόν σε σχέση με το ΜΕΚ και επίσης είναι διατηρημένη η Κομισιόν να, να συμπεριλάβει αυτή τη διάσταση ότι θα πρέπει σε πρώτη φάση τουλάχιστον να εξαντλούνται ε, τα εθνικά μέσα. Κύριος Μπούχνα, η Κομισιόν είναι διατεθειμένη να υπογράψει συνθήκη, συμφωνία, που θα περιλαμβάνει σοβαρά κεφάλαια που θα αφορούν τις επενδύσεις και το εμπόριο. Και όταν λέω σοβαρά εννοώ να προβλέπονται και συγκεκριμένοι μηχανισμοί κυρώσεων. Δεύτερο ερώτημα. Τι συμβαίνει με τα γενώσιμα φάρμακα. Στο παρελθόν είχαμε αντιμετωπίσει σοβαρότατα προβλήματα θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω την Κομισιόν ε, πώς σκοπεύει να χειριστεί το συγκεκριμένο θέμα. Η κυρία Χάιντι Χάουταλα. Ευχαριστώ. Οι πρόεδροι Τούσκ, Γιούγκερ και η κυρία Μογκερίνη έχουν ε, επισημάνει ε, το, τη σημασία του θέματος της απουσίας διακρίσεων στην Ινδία. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω την πρέσβυρα. Πώς χειρίζεται τα ζητήματα ε, των διακρίσεων ε, σε σχέση με ε, των διακρίσεων που δέχονται πληθυσμιακές ομάδες που δεν ανήκουν σε κάστες στην Ινδία γιατί είναι ένα θέμα που επηρεάζει και τις διεθνείς μας σχέσεις. κυρία Πρέσβυρα, ε, ήταν μια ερώτηση για εσάς, που απευθυνόταν σε εσά. Θέλετε να απαντήσετε. Η απάντηση είναι πολύ απλή οι αρχές μας παραδόσεις αλλά και το σύνδειγμα μας και οι νόμοι μας με ολοκληρωμένο τρόπο προβλέπουν την αντιμετώπιση και την καταπολέμηση οποιασδήποτε διάκρισης βάσει κάστας, φύλου, θρησκείας. Προφανώς σε μια χώρα 1,3 ε, δισεκατομμυρίων ε, πολιτών φαινόμενα εμφανίζονται καθημερινά. Αλλά το σημαντικό είναι ότι κάθε πολίτης μας έχει το δικαίωμα να προσφεύγει σε, στην ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Θεωρούμε ότι έχουμε επαρκείς μηχανισμούς προκειμένου να αντιμετωπίζεται το θέμα. Είναι ένα εσωτερικό μας θέμα, το οποίο βεβαίως και ε, εξετάζουμε και προσπαθούμε να λύσουμε. Και τον Αύγουστο μάλιστα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνώρισε τις ε, εν λόγω προϋπος ε, προσπάθειες της Ινδίας. Εγώ δεν θα αρνηθώ ποτέ ότι τέτοιου είδου φαινόμενα εμφανίζονται κάθε μέρα. Αλλά σε μια χώρα με τον πληθυσμό της δικής μας, με 29 κρατήδια, καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να υπάρξει μια ολοκληρωμένη, εξειδικευμένη αντιμετώπιση του θέματος. Εκτιμούμε βέβαια στο γεγονό ότι ε, σας απασχολεί το θέμα και ευχαριστούμε για τη συγκεκριμένη παρέμβαση. Ευχαριστώ πολύ κυρία Κιόνιχ για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Ε, μιλάω συχνά γρήγορα. Ελπίζω οι διερμηνείς να μπορούν να με ακολουθήσουν. Να ξεκινήσω με ένα σχόλιο. Όπω είπε και η κυρία Πρέσβυρα, υπάρχουν κάποιε προκαταρκτικέ διαπραγματεύσει, οι οποίε θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι διαρευνητικού χαρακτήρα, προκειμένου να δούμε πού βρίσκεται η κάθε πλευρά. Και με αυτό να περάσω στο πρώτο θέμα. Αυτό που προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε είναι ότι ό,τι και αν τεθεί τελικά επιτάπητο, προκειμένου να συζητηθεί φέτο, θα πρέπει να είναι τέτοια φύση ώστε να έχουν όλοι πλήρη αντίληψη των δυνατοτήτων αλλά και των περιορισμών. Αυτό νομίζω ότι είναι απόλυτη προϋπόθεση, ελάχιστη προϋπόθεση προκειμένου να ξεκινήσουν αλλά και να ολοκληρωθούν αυτές οι διαπραγματεύσεις Γιατί αυτό που μας εμποδίζει αυτή τη στιγμή είναι το γεγονός ότι έχουμε και από τις δύο πλευρές πολύ ψηλέ προσδοκίε και δεν έχουμε συζητήσει επαρκώς το, το ζήτημα της ευελιξίας που μπορεί να επιδείξει ο καθένας. Ε, γι' αυτό και άλλωστε οι διαπραγματεύσεις είχαν, είχαν σταματήσει το 2013, αλλά όπως είπα ο, ο, ο καιρός πέρασε και πρέπει πλέον να δούμε, να κάνουμε ένα απολογισμό, να δούμε πού ακριβώς βρισκόμαστε σήμερα πια. Επενδύσεις. Ε, αναφέρθηκα και στην παρουσίασή μου ότι η Ινδία επιμένει στο να συμπεριληφθεί το θέμα των επενδύσεων στην ε, συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών. Βεβαίω, μετά την απόφαση του δικαστηρίου, εγώ δεν μπορώ να σα πω ότι θα εγκαταλείψουμε τη συγκεκριμένη στάση. Σίγουρα θα συζητήσουμε το ζήτημα τη προστασία των επενδυτών από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και το, νέο ε, πρότυπο BIT που έχει προτείνει η Ινδία. Τώρα το ποια θα είναι η στάση μας είναι πολύ πρόημο να σας το πω αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι σημαντικό είναι αυτή τη στιγμή να επικεντρωθούμε στο ποιε ακριβώς είναι οι επιδιώξεις μας και είναι οι στόχοι μας και από τις δύο πλευρές προκειμένου να δούμε αν μπορούμε να συμφωνήσουμε. Για, την, ε, για, τα, για τα μέσα ε, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην υπάρχει μια συσσόρευση υπερβολικά πολλών ε, εθνικών ε, ε, ένδικων μέσων, να μην καθυστερεί δηλαδή η διαδικασία απόδοσης, απονομής δικαιοσύνης. Και αυτό είναι ένα θέμα που μας ενδιαφέρει πολύ, γιατί θέλουμε να υπάρχει η δυνατότητα και να, να, να καταλήγουν κάπου οι διαφορές στον τομέα των επενδύσεων, όταν αυτές θα ανακύπτουν. Για την εντολή. Εγώ προφανώς δεν μπορώ να σχολιάσω είναι απόφαση του, του Συμβουλίου να δημοσιεύσει τη συγκεκριμένη εντολή. Η Κομισιόν έχει ξεκαθαρίσει την πρόθεσή της ότι θέλει να δημοσιεύονται στο εξή όλες οι εντολές που αποφασίζει το Συμβούλιο και νομίζω ότι αν κινηθούμε σε αυτή τη δικαδέστηση θετικό θα είναι. Για το TST. Είναι ένα από τα κεφάλαια τα οποία έχουν συζητηθεί επί μακρόν αλλά εξακολουθούμε να εμ, χρειαζόμαστε και περαιτέρω συζητήσει. Γιατί το, το, θέμα είναι ακαθόδε. Έχουμε πολύ ψηλέ φιλοδοξίε σε αυτό το θέμα. Ε, εμείς, ε, ε, εμείς ε, έχουμε διαπιστώσει ότι οι Ινδοί παραδοσιακά δεν εντάσσουν το συγκεκριμένο κεφάλαιο στις δικές τους συμφωνίες που υπογράφουν με οργανώσεις και άλλα κράτη αλλά όπως και με άλλους εταίρους μας, ε, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας πω ότι έχει συμφωνηθεί ένας μηχανισμός επιβολής κυρώσεων, γιατί όπως συζητήσαμε στο προηγούμενο θέμα για το Μεξικό, δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί ε, οι σχετικές διαβουλεύσεις εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο το, δικό μα. Μόλι όμω ολοκληρωθούν, βεβαίω θα μπορέσουμε να διαμορφώσουμε τη στάση μα και θα σα ενημερώσουμε σχετικά. Προφανώ δεν θα πετάξουμε στα σκουπίδια όλα όσα έχουμε επιτύχει μέχρι στιγμή, αλλά βεβαίω πρέπει να υπάρξει μια επανέναρξη των συζητήσεων και να δούμε και ορισμένα θέματα από την αρχή. Βεβαίω είναι σημαντικό το ζήτημα τη ευελιξία που, ε, που, που δίνεται στο πλαίσιο του ΠΟΕ για τα φάρμακα. Και εδώ έχουμε επιδείξει προσήλωση στι διαπραγματεύσει μα με του Ινδού και δεν, δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε ούτε αυτή τη φορά. Γιατί καταλαβαίνουμε πόσο, είναι, πόσο σημαντική είναι η βιομηχανία των γενώσιμων φαρμάκων, όχι μόνο στην Ινδία, αλλά σε ολόκληρο τον αναπτυσσόμενο κόσμο. Ε, Επίση, δεν συζητούμε σε καμία περίπτωση μείωση των προτύπων για την ασφάλεια των τροφίμων και για τις ε, ε, υπηρεσίες. Ε, βεβαίως ε, ο, ο τρόπος που προσκυγούμε το ζήτημα αυτό χαρακτηρίζεται κυρίως από το Modifor. Ε, κύριε Κάμπελ, θέλετε να ολοκληρώσετε τη συζήτηση αυτή με μια τελευταία πρόταση. Εγώ, κύριε Πρόεδρε, θα μπορούσα να να συντάξω και μια ολόκληρη έκθεση, αν θέλετε, και μάλιστα και με το πλήρες όνομα μου, Κάμπελ Μπάνερμαν. Ωραία, πάμε στις ψηφοφορίες λοιπόν, λέει ο πρόεδρο. Και θα ξεκινήσουμε με μια δοκιμαστική ψηφοφορία, όπως πάντοτε, για να δούμε αν λειτουργούν τα συστήματά μας, αν έχουν όλοι τις κάρτες τους. Παρακαλώ, ψηφίστε για να δούμε αν λειτουργούν όλα σωστά. And the vote is closed. Πέρασε Πέρας ψηφοφορίας. Okay. Good. Everything is fi fixed and then we came uh, we come to... Ωραία. Λειτουργούν τα πάντα. Μια χαρά. Πάμε, περνάμε στην πρώτη ψηφοφορία. Πρώτη ψηφοφορία για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο dumping. Να ψηφίσουμε παρακαλώ. And the vote is closed. Πέρας της προφορίας. Εγκρίνεται με ευρία πλειοψηφία. Συγχαρητήρια στον κύριο Φιέλνε, τον συγκητή μας. Επόμενο θέμα. Σημείο 16 γνωμοδότηση για τη μεταρρύθμιση του συστήματος των ιδίων πόρων τη ευρωπαϊκή Ένωση, Ο κ. Φαντεκάμ είναι ο συντάκτη αυτής τη γνωμοδότηση. Πρώτον, ε, συμβαστική τροπολογία 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 1. Όχι, όχι, καταπίπτει, συγγνώμη. Τροπολογία 2. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 9 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 13 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 18 υπέρ κατά ας το ξανακάνουμε λίγο υπέρ κατά αποχές θα το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ για να είμαστε σίγουροι. And the vote Πέρα τη ψηφοφορία, απορρίπτεται. Συμβαστική 5 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Okay. Okay. So this amendment 19, we will have be in mind because we will. But it falls. It was just a mistake of renumbering. Oh, it was a response. Okay. So. Ωραία. Τροπολογία 27 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ, κατά, αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά καλύτερα να το ελέγξουμε. Άρχισε η ψηφοφορία, ψηφίστε παρακαλώ. And the closed. Πέρας. Ναι, απορρίπτεται. Then we have και περνάμε στη συμβαστική 8. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 35. I have to include the last compromise last minute. So next time, please uh, try to renumber the correct. Uh, so. Και περνάμε στην τελική ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Er, er ναι, υπήρξε ένα πρόβλημα με την αρρύθμιση των ε, τροπολογιών. Γι' αυτό αργήσαμε λίγο εδώ στο τέλος, αλλά περνάμε τώρα στην ε, τελική ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. And the vote is closed. Πέρας ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κύριε Βαντεκάμπ. Εδώ δεν είναι. Όχι. Δεν πειράζει. Και σημείο 17. Συστάσεις προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΕ. σχετικά με τις απομονωτές για τη Συνολική Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Αζερβαϊτζάν. Έχουμε κάποιες τροπολογίες του κύριου Τάκ Υπάρχει πρόταση να ψηφιστούν από κοινού. Δεν βλέπω να υπάρχει αντίρρηση. Ποιο είναι υπέρ των τροπολογιών 1 έως 19. Κατά, αποχές, εγκρίνονται. Και τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. And the vote is closed. Πέρας Εγκρίνεται. Με μεγάλη πλειοψηφία. Ευχαριστώ. Αυτή ήταν η πολύ σύντομη ψηφοφορία που είχαμε για σήμερα το πρωί. Αν θέλετε να εγκαταλείψετε την αίθουσα, κάντε το, σας παρακαλώ, αλλά ησύχως. Και περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης Dann kommen wir zu Punkt 18 und 19. Σημεία 18 και 19 που αφορούν τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου αφενός το ζήτημα της ε, έκθεσης της αποστολής που συμμετείχε στην υπουργική διάσκεψη του ΠΟΕ στον Πουένος Αέρος αλλά και γενικά ε, ποιο θα είναι το μέλλον του ΠΟΕ. Γιατί γνωρίζουμε όλοι ότι το αποτέλεσμα της διάσκεψης στον Buenos Aires ήταν απογοητευτικό και αμφισβητήθηκε για πρώτη φορά στα σοβαρά ο τρόπος λειτουργίας του ΠΟΕ. Η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποτελούν από 14 μέλη. Συμμετείχε λοιπόν στην ετήσια υπουργική διάσκεψη και στις προκαταρκτικές συναντήσεις και στην ίδια την υπουργική διάσκεψη και βεβαίως σε μια σειρά από διμερείς συναντήσεις με διάφορους υπουργούς του, της Ιαπωνίας για παράδειγμα, της Αυστραλίας ε, και της Αργεντινής. Από αυτή την άποψη ήταν πολλά υποσχόμενη η επίσκεψη της αντιπροσωπείας μας. Ωστόσο, η κοινοβουλευτική διάσκεψη, η διοικούσα επιτροπή δηλαδή της ε, κοινοβουλευτικής διάσκεψης, συζήτησε, συζήτησε επί μακρόν ένα έγγραφο το οποίο επρόκειτο να δημοσιευθεί στο τέλος καταλήξαν τελικά σε ένα τέτοιο έγγραφο, το οποίο όμως δεν έχει κανένα ουσιαστικό περιεχόμενο. Διότι δεν κατέστη δυνατόν να καταλήξουμε σε έναν επικοδομητικό συμβιβασμό. Η, το πρόβλημα δημιουργήθηκε ιδίως από μία χώρα, την Ινδία, η οποία μπλόκαρε πολλά από τα θέματα, θέματα της ε, διεθνούς εμπορικής πολιτικής. Μόνο για ένα θέμα ενδιαφέρθηκε η Ινδία, που αφορούσε την αποθήκευση και την ασφάλεια των ε, τροφίμων. Αυτό ήταν διατεθειμένοι να το συζητήσουν, αλλά όλα τα, όλα τα άλλα όχι. Και έτσι οδηγήθηκαν σε μια κατάσταση όπου σε όλους τους άλλους τομείς δεν καταφέραμε να επιτύχουμε κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα πρέπει πραγματικά να δούμε τι θα κάνουμε στο μέλλον με αυτή την κοινοβουλευτική διάσκεψη. Προσωπικά θεωρώ ότι δεν έχει κανένα νόημα να συγκεντρώνονται βουλευτές από όλο τον πλανήτη σε, ένα, σε μια συγκεκριμένη χώρα, σε μια συγκεκριμένη πόλη, να συζητούν δύο μέρες και τελικά να καταλήγουν σε ένα έγγραφο το οποίο ούτε το γνωρίζει κανείς, αλλά ούτε έχει και κανένα ε, ουσιαστικό περιεχόμενο. Στο επίπεδο της ε, υπουργικής διάσκεψης μάλιστα ρωτήθηκαν πολλοί υπουργοί που συμμετείχαν αν ξέρουν ε, για την ύπαρξη αυτού του εγγράφου της κοινοβουλευτικής διάσκεψης και η απάντηση ήταν πάντοτε όχι. Ε, αυτό δεν έχει νόημα. Εγώ θα έλεγα ότι πρέπει να ενισχύσουμε την κοινοβουλευτική διάσταση, γιατί ακριβώ αυτό είναι και ο ρόλο μα. Θέλουμε ω βουλευτέ να προωθήσουμε και να ενισχύσουμε τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Αλλά αν έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση όπου ε, δεν υπάρχει καμία δυνατότητα να επιτυχάνει κανεί ορατά, απτά αποτελέσματα, ε, τότε δεν έχει νόημα να την ακολουθεί αυτή τη διαδικασία. Συζητήσαμε το θέμα αυτό και στην ε, ε Διευθύνουσα Επιτροπή, εδώ σε επίπεδο ε, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και καταλήξαμε στο να θεσπίσουμε, να καταρτήσουμε μια, ε, μια σειρά από προτάσεις τις οποίες θα υποβάλουμε και στην κοινοβουλευτική διάσκεψη του ΠΟΕ θα τη διανύμουμε βεβαίω και στους εταίρους μας, σε όλους τους συμμετέχοντες, σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες, ώστε στην επόμενη συνάντηση, συνάντηση του Μαρτίου να μπορέσουμε να συζητήσουμε αυτές τις προτάσεις ρύθμισή μας, με απότερο στόχο, όπως είπα, να επαναπροσδώσουμε κάποιο νόημα στη διαδικασία της κοινοβουλευτικής διάσκεψης. Δεύτερον, Βεβαίω, ε, υπήρξε ε, και πραγματοποιήθηκε η ενδέκατη υπουργική διάσκεψη ΠΟΕ. Εκεί μάλιστα δεν καταλήξανε ούτε καν σε έγγραφο. Βεβαίως οι ελπίδες ήταν περιορισμένες ως προς το τι θα μπορούσε να επιτευχθεί. Συζητήθηκε για παράδειγμα το ζήτημα της απαγόρευσης ε, των επιδοτήσεων στην Αλία και αν και κατά πόσο ένα τέτοιο στόχος θα μπορούσε να είναι εφικτός με ε, σκοπό την ενίσχυση της βιωσιμότητας της αλληλείας. Υπήρξαν κάποιες συζητήσει για κάποιες ε, υπηρεσίες, για το ηλεκτρονικό εμπόριο για παράδειγμα. Συζητήθηκαν όλα αυτά τα θέματα χωρίς όμως να καταλήξουμε σε τίποτα. Ούτε καν ως προς τα επόμενα βήματα που θα αναλυθούν. Με αποτέλεσμα να έχουμε μπροστά μας το ενδεχόμενο και την πιθανότητα σύναψης διμερών συμφωνιών ή πολυμερών αλλά μόνο μεταξύ συγκεκριμένων ομάδων χωρών. Κάτι που απέχει βεβαίως από μια παραδοσιακή και κλασική πολυμερή προσέγγιση. Και όλα αυτά νομίζω ότι μας οδηγούν στην ανάγκη να ε, συζητηθεί και το μέλλον του ΠΟΕ. Δύο χρόνια προετοιμάζαμε αυτές τις διασκέψεις. Τρεις χιλιάδες άνθρωποι πήγαν στον Buenos Aires. Ε, από μια τέτοια τεράστια διαδικασία, χρονοβόρα και δαπανηρή, να μην βγαίνει τίποτα, ούτε καν ένα έγγραφα, ε, τότε νομίζω ότι δεν μπορούμε να αποφύγουμε το ερώτημα κατά πόσο έχει νόημα. Και νομίζω ότι εναπόκειται και σε εμά ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να βάλουμε μπρο τι μηχανέ και να διερευνήσουμε αλλά και να αξιοποιήσουμε κάθε δυνατότητα προκειμένου να τονώσουμε τη διαδικασία αυτή, να τη μεταρρυθμίσουμε με στόχο να διατηρηθεί βεβαίως το σύστημα αυτό. Εγώ δεν λέω ότι δεν είναι ε, σημαντικό το να υπάρχει ε, ο ΠΟΕ και εμάς ως Ευρωπαϊκή Ένωση μας ενδιαφέρει και μας συμφέρει πολύ να υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες για το διεθνές εμπόριο. Αυτά εισηγητικά από εμένα θα ήθελα να δώσω το λόγο τώρα στα μέλη της αποστολής που συμμετείχαν η κυρία Μαγκίνες, ο κύριος Βίνκλερ, δεν είναι κανείς τους εδώ. Ίνμα, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. <clears throat> Η εισαγωγή σας ήταν τέλεια, συγκεκριμένη, πλήρης και ενδελεχής. Ούτως ή άλλως πρέπει να κάνουμε αυτή την ανάλυση αυτών τον προβληματισμό. Τι θέλουμε από τον ΠΟΕ, πώς θέλουμε να λειτουργήσει ο ΠΟΕ, η κοινοβουλευτική του συνέλευση και τι μηχανισμούς μεταρρύθμισης θα πρέπει να εξετάσουμε. Πέρα από το αποτέλεσμα που ήταν ολέθριο, όπως το εξήγησε πολύ ωραία ο Πρόεδρος, πρέπει να διδαχθούμε ε, για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τα πράγματα, ε, να τα διορθώσουμε, ε, να σκεφτούμε τι έγινε για να τα αλλάξουμε. Είναι πολύ σημαντικό ότι υπήρχε λίγο ενδιαφέρον για το έγγραφο το οποίο εγκρίναμε σε σχέση με το περιεχόμενό του. Γι' αυτό θα έπρεπε να κάνουμε μία πρώτερη εργασία με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, με τις ΜΚΟ, με τους ε, οικονομικούς και κοινωνικούς φορείς, ούτως ώστε να αισθανθούν ότι τους ενδιαφέρει αυτό το πράγμα, ότι είναι δική τους υπόθεση. Ειδικά η Κοινοβουλευτική Συνέλευση και η Υπουργική Σύνοδος. Μην ξεχνάτε ότι οι δημαγωγοί, οι λαϊκιστές, ε, η δεξιά με τον προστατευτισμό της, ξέρετε πολύ καλά ότι είναι κατά της, του, του πολυμερού συστήματος, της παγκοσμιοποίησης, είναι υπέρ των ακραίων εθνικισμών κτλ. Ε, μην ξεχνάτε όμως ότι υπάρχουν πολλά κόμματα που είναι υπέρ της πολυμέρειας, του πολυμερού συστήματος. Ε, και μέσα στα στους φορείς αυτούς που υπάρχει αντίθεση, θα πρέπει να βρούμε ε, στοιχεία για να βασιστούμε σε αυτά, για να προσερκίσουμε και άλλους. Νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι σε θέση να παίξει ένα ρόλο έτσι, ηγετικό, να κάνει προτάσεις ε, για να αισθανθούν και οι υπόλοιποι ότι τους αφορά αυτή η ιστορία. Είναι σημαντική να γίνει αυτή η ανάλυση, αυτή η συζήτηση και να υπάρξουν συγκεκριμένες προτάσεις. Ευχαριστώ. Ο David Μάρτιν. Ευχαριστώ. Φυσικά συμφωνώ απόλυτα με, με εσά ότι υπήρχαν απογοητευτικά αποτελέσματα από την ε, εκδήλωση. Τρεις φάσεις ε, είδαμε. Πριν πάμε στην Υπουργική, ήταν η δήλωση του Buenos Aires δεν θα πρέπει να υποτιμούμε το γεγονός ότι οι λατινοαμερικανικές χώρες, ε, επειδή ακριβώς η διάσκεψη έγινε στο Buenos Aires, ε, διάφοροι πρόεδροι λατινοαμερικανικών χωρών ήταν υπέρ ε, του συστήματος του ΠΟΕ, του πολυμερού συστήματος. Είναι θετικό το ότι οι πρόεδροι διαφόρων λατινοαμερικανικών χωρών, τεσσάρων λατινοαμερικανικών χωρών, τάχθηκαν υπέρ. Δέκα χώρες ε, προσυπέγραψαν υπέρ ε, και είναι σημαντικό να κάνουμε περισσότερα για να ενθαρρύνουμε και το ρόλο των ε, γυναικών. Πέρα από, την, από όλα αυτά, για την κοινοβουλευτική συνέλευση συμφωνώ με την αξιολόγησή σας. Ε, δυστυχώς μαζί με τα ξερά πετάξαμε και τα χλωρά. Ε, το θέμα είναι πώς θα βρούμε τρόπους για να μεταρρυθμίσουμε αυτό είναι το βασικό στοιχείο, γιατί έχει νόημα οι βουλευτές από όλο τον κόσμο να συνέρχονται, να συζητάνε. Ε, πρέπει να υπάρχει κοινοβουλευτικό έλεγχος στον ΠΟΕ, πρέπει να συνεχίσουμε. Δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν το κάναμε. Για την Υπουργική δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά. Πρέπει να αναγνωρίσουμε πάντως ότι είναι πολύ δύσκολες εποχές τώρα αυτές ε, και ασυνήθιστες. Δεν θα έλεγα αντίθεση, αλλά θα έλεγα σχεδόν ότι δεν συμμετέχουν οι Αμερικάνοι ας πούμε, στη διαδικασία, δεν έχουν καμία διάθεση για να δεσμευτούν και αυτό δεν βοήθησε το γεγονός ότι δυσκολε... υπάρχει δυσκολία και γενικά με την παγκόσμια οικονομία. Ε, αυτό οδήγησε σε απογοητευτική κατάσταση στην Υπουργική. Αυτό παρόλα αυτά ε, δεν θα πρέπει να μας κατεβάσουμε τα χέρια. Ο Πολ Ρούμπι, ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω, να σας ευχαριστήσω, γιατί αυτή η διάσκεψη δείχνει πόσο δύσκολο είναι να συνέλθουμε ε, τόσες χώρες για να βρούμε ένα κοινό πλαίσιο. 160 χώρες. Ε, άτομα έχουν ε, βέτο και μπορούν να μπλοκάρουν ε, την πορεία προς τα εμπρός και να, μην, και να μπλοκάρουν μάλιστα και τη σύνταξη συμπερασμάτων. Όχι μόνο στην Υπουργική Σύνοδο, αλλά και στη συνεργασία μας με τον ΠΟΕ πρέπει να υπάρξει μεταρρύθμιση. Τώρα, για την κοινοβουλευτική διάσκεψη. Ξεκινάμε από εκεί για να αναπτύξουμε περαιτέρω το πλαίσιο της συνεργασίας. Είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι οι βουλευτές ενημερώνονται όπως και οι υπουργοί στο τέλος των διαπραγματεύσεων. Ίσως θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει πιο τακτική ενημέρωσή του όμω, όχι μόνο στο τέλος, για να υπάρχει πραγματική ισοτιμία με τους υπουργού. Θα πρέπει να ξαναδούμε τους στόχους που θέλουμε να πετύχουμε. Υπάρχει, υπάρχει ο, ο στόχος της βιώσιμης ανάπτυξης. Δεν το συζητήσαμε πολύ κατά τη διάρκεια Υπάρχει το θέμα της ανάπτυξης παγκόσμιας στρατηγικής Αυτό που με εντυπωσίασε πιο πολύ είναι ότι δεν υπήρξε καμία συνένεση ούτε σε επίπεδο υπουργών, ούτε σε επίπεδο βουλευτών. Και έτσι δεν καταλήξαμε συμφωνία. Θα πρέπει να βρούμε άλλη προσέγγιση λοιπόν από αυτήν. Θα πρέπει να ασχοληθούμε περισσότερο με τους ε, μηχανισμούς επίλυσης ε, διαφορών. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, λέει η κυρία Μακλάρκιν. Ήταν ε, απογοητευτικό σε πολυμερές επίπεδο το αποτέλεσμα, αλλά γίνονται και άλλες εργασίες αναφέρθηκαν από τους διαπραγματευτές για τη συμφωνία με το Μεξικό και το Μεκοσούρ παράπλευρα, στα πλαίσια αυτών των διαπραγματεύσεων του ΠΟΕ, έγιναν καλές επαφές με τους άλλους. Είχαμε καλές επαφές με την Αυστραλία ε, και με τους Αργεντινούς. Έγιναν καλές συζητήσεις και μπορούμε να βασιστούμε σε αυτές. Στην ε, κοινοβουλευτική διάσκεψη, εγώ και ο συνάδελφος κάναμε μία σύνοδο για το ηλεκτρονικό εμπόριο και για την ε, παγκόσμια διάσταση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ήταν μια πολύ έντονη έτσι, συζήτηση και είχαμε ερωταποκρίσεις που κράτησαν πάνω από μία ώρα. Ε, κάποιες ήταν πιο θετικές, υπήρχαν αντιδράσεις, ε, έγιναν συζητήσεις και με αφρικανικές χώρες και με την Ινδία για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Ο ρόλος μας ε, σε αυτή την κοινοβουλευτική διάσκεψη είναι να επηρεάσουμε και να κάνουμε αυτές τις συζητήσεις και να ενημερώσουμε τον κόσμο, ούτω ώστε να πιστούν και άλλοι βουλευτές για να πιέσουν να υπάρξουν ε, συζητήσεις ε, για άλλα θέματα σε πολυμερές επίπεδο. Ε, π.χ. ηλεκτρονικό εμπόριο στο μέλλον. Κρίμα που δεν πετύχαμε κάτι παραπάνω. Οι συζητήσεις που είχαμε στις συνεδριάσεις πιστεύω ότι θα παίξουν κάποιο ρόλο, θα αποτελέσουν μια βάση ούτω ώστε να υπάρξει πρόοδος στο μέλλον. Ευχαριστώ, λέει ο κ. Κάμπελ. Ε, να προσθέσω κι εγώ ε, ότι ναι, είμαστε απογοητευμένοι για το τελικό αποτέλεσμα της Υπουργικής Διάσκεψης. Ε, εγώ δεν είχα παραστεί πριν, ε, που δεν είχα παραστεί πριν. Ήταν εντυπωσιακό το γεγονό ότι εμφανίστηκαν τόσε πολλέ χώρε. Δεν κατάρρισε καμία χώρα. Ήταν όλε παρούσε, αλλά δεν ήθελαν να δεσμευτούν. Όπω η Ινδία, η Κίνα και η ΙΠΑ δεν βοηθούσαν με τη στάση του στη διαδικασία. Ε, δυστυχώς. Το επίγον θέμα είναι ότι υπάρχει έλλειψη μελών ε, στα πάνελ. Δεν μιλάω για τους δικαστές, μιλάω για τους, ε, τα μέλη του πάνελ. Ε, είναι ευαίσθητο θέμα και υπάρχει ένα πρόβλημα με τον ε, μηχανισμό επίλυσης διαφορών. Είχαμε την ανακοίνωση από πλευράς Αμερικανών για τα, τους δασμούς, για τις κορεάτικες, τα κορεάτικα πλυντήρια και τα κινέζικα φωτοβολταϊκά ε, κάποια στιγμή θα υπάρξει α, μια κρίση και όλο το σύστημα θα, θα αμφισβητηθεί έτσι. Ε, είναι σοβαρό θέμα. Τέλος. Η κοινοβουλευτική διάσταση είναι πολύ σημαντική. Το γεγονός ότι συζητάμε για το εμπόριο, ότι υπάρχουν ε, άνθρωποι από όλο τον κόσμο, από το ας πούμε αργεντίνικο κοινοβούλιο, καθώς και οι διμερείς επαφές που είπε η ΕΜΑ, ήταν πολύ χρήσιμες. Είναι πολύ σημαντικές και βοηθάνε πάρα πολύ αυτές οι διμερείς. Και Ευχαριστώ την ε, ομάδα που οργάνωσε αυτές τις επαφές. Η κυρία Χάουταλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την πολύ εκτεταμένη έκθεση, ή ε, μάλλον παρουσίαση. Για τους πράσινους, το θέμα της εφαρμογής των κανόνων είναι θέμα κλειδί. Και πιστεύω, όπως και οι προλαλήσαντες, ότι είναι πολύ σημαντικό να βρεθεί μια λύση στο μηχανισμό επίλυσης διαφορών σε αυτό το θέμα. Γιατί εάν δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ε, εφαρμογή των κανόνων του ΠΟΕ, τότε πώς μπορούμε να πιστεύουμε ότι η οργάνωση θα εξασφαλίσει νέους κανόνες ας πούμε, για το ηλεκτρονικό εμπόριο ή για οτιδήποτε άλλο. Είναι άδικο που μπλοκάρει η Αμερική την, το διορισμό μελών του Σώματος Προσφυγών η κριτική των ε, Αμερικανών για το μηχανισμό επίλυσης διαφορών πρέπει να πούμε ότι έχει, έχει κάποια βάση, έτσι. Και θα πρέπει, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να το συζητήσουμε το θέμα αυτό. Επίσης, θα ήθελα να σας πω ότι η διαβούλευση ή μάλλον ε, έχουμε από τη μία τον ΠΟΕ και από την άλλη την ατζέντα του ΟΗΕ για τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Αυτά δύο πάνε παράλληλα και θα πρέπει να ενισχύσουμε το διάλογο μεταξύ του ΠΟΕ και του ΟΗΕ. Θα έλεγα μάλιστα και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Να βάλω και την Παγκόσμια Τράπεζα στην εξίσωση. Και ίσως η Επιτροπή μας θα μπορούσε να προωθήσει έτσι, το διάλογο αυτό ε, από διάφορες οργανώσεις να τους καλέσουμε ας πούμε, για να δούμε πώς μπορεί να γίνει. Είναι μια πιο γενική ε, παρατήρηση. Δεν έχουμε ένα μηχανισμό που, θα, που εξετάζει πλήρως την εφαρμογή των στόχων του 2030. Και αυτό αφορά γενικά ε, το εμπόριο, αλλά όχι μόνο. Υπάρχει, υπάρχουν και άλλα θέματα. Το εμπόριο είναι κομβική σημασία. Φυσικά ε, σκεφτόμαστε ως Επιτροπή ποιο είναι το αποτέλεσμα της σημαντικής αυτής διάσκεψης προβληματιζόμαστε. Αυτές ήταν οι... Και τώρα θέλουμε να ακούσουμε και τις παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σημειώσαμε τις απόψεις που εκφράστηκαν σήμερα και θα ενημερώσουμε τη δική μας ε, ομάδα της Κομισιόν για τη στραγική ε, τη μετέπειτα στρατηγική. Είμαστε σε πρώιμη φάση, θα πάρει χρόνο το θέμα, όπως και άλλα μέλη του ΠΟΕ, απλώς ακόμα σκεφτόμαστε τους λόγους, τους υποκείμενους λόγους ε, για τους οποίους ε, η συζήτηση στον ΠΟΕ ήταν αυτή που ήταν, που ήταν και έδωσε αυτό το απογοητευτικό αποτέλεσμα. Να σας πω σε αυτή τη φάση ότι η αξιολόγησή μας για το που βρισκόμαστε συγκλίνει γενικά με τις απόψεις και τα αισθήματα που ακούστηκαν σήμερα εδώ πήγαμε στην MC11 ε, με ανοιχτά τα μάτια, υπήρχαν δυσκολίες με τη λειτουργία της διαπραγμάτευσης, είχαμε και νέα προβλήματα, υψηλό επίπεδο αβεβαιότητας, ε, κυρίως ε, μεταξύ άλλων λόγω της στάσης της κυβέρνησης των Αμερικανών, οι οποίοι μπλόκαραν, ας πούμε, την, διάφορα πράγματα, ακόμα και τη συνήθη διεκπαιρέωση υποθέσεων από τον ΠΟΕ σε διάφορα επίπεδα ήταν αρνητική η στάση τους και επίσης δεν υπήρχε και πολιτική ηγεσία, ας πούμε, που θα στήριζε το σύστημα. Νομίζω ότι να υπάρξει πολιτική στήριξη και ηγεσία θα, χρειαζόταν. Ε, και αυτό που κάνουν οι βουλευτές στον ΠΟΕ είναι πολύ χρήσιμο και εκ των όνων κάνε ώστε να κρατήσουμε την εστίαση ε, στον ΠΟΕ οι πιθανότητες επιτυχίας ήταν ε, ισχνές. Εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να αυξήσουμε αυτές τις πιθανότητες επιτυχίας. Ε, εμείς κάναμε συγκεκριμένες προτάσεις, τις βάζαμε στο τραπέζι. Αυτό κάναμε ούτως ή άλλως όλο το 17. Ούτως ή άλλως ένα μέλος με αυτόν τον τρόπο ασκεί ηγετικό ρόλο, ε, με το να προτείνει συγκεκριμένα πράγματα. Δυστυχώς όμως ε, η απογοήτευση ήταν δεδομένη. Όταν δεν μπορούσαμε να πετύχουμε τίποτα για τη γεωργία ε, και αυτό οδήγησε σε μια επίπτωση ντόμινο, ας πούμε, που επηρέασε όλα τα υπόλοιπα θέματα που ήταν υπό συζήτηση στη διάσκεψη. Ως αποτέλεσμα και η υπουργική διάσκεψη δεν συμφώνησε ούτε, μία, ούτε επί μιας υπουργικής δήλωσης, που θα ήταν η βάση για, κάπως για να προχωρήσουμε. Ε, επομένως, έχουμε αβεβαιότητα για το τι θα κάνουμε τώρα και κατά την άποψή μας ενισχύει την ανάγκη για να διευρύνουμε την προσέγγισή μας, να υπάρξει μεγαλύτερη ευελιξία, ε, να βρούμε τρόπους για να την εξασφαλίσουμε στην διαπραγματευτική εντολή. Αυτό θα είναι το θέμα μας στους επόμενους μήνες με τα μέλη του ΠΟΕ. Τώρα, για το πολυμερές επίπεδο, διάφορες κοινέ δηλώσεις όντως συμφωνήθηκαν ε, μερικές φορές και από πολλά μέλη που θα αποτελέσουν αυτές μια απαρχή συζητήσεων. Εμείς θα συζητήσουμε μαζί με τους υπόλοιπους, ούτω ώστε να μείνει ανοιχτή η πρωτοβουλία και να, και να είμαστε προσκολλημένοι στο σύστημα του ΠΟΕ. Σε πολυμερές επίπεδο θα ξαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις για τις επιδοτήσεις. Είναι ένα σημείο στην ατζέντα που συμφωνεί με μία εντολή πέρα από την εντολή που έχει ο ΠΟΕ και έχει να κάνει με την εντολή που υπάρχει για τους στόχους της χιλιετίας, όπως είπε και η κυρία Χαουτάλα, τους βιώσιμους στόχους της χιλιετίας. Ε, τους επόμενους μήνες θα ασχοληθούμε όχι με τη διαπραγματευτική εντολή, όσο με την ε, τακτική λειτουργία του ΠΟΕ, τη θεσμική του λειτουργία και το θεσμικό του ρόλο που θα πρέπει να διατηρήσουμε. Επίσης θα ασχοληθούμε ενεργά με ε, μια, ένα δεύτερο μεγάλο μέλημα στον ΠΟΕ, που είναι τι γίνεται, με το βραχείο επίλυσης διαφορών ε, και με το θέμα του σώματος προσφυγών. Ε, η Κομισιόν και η Επίτροπος ε, Μάστον θεωρεί ότι το σώμα προσφυγών αποτελεί μεγάλο κίνδυνο για το σύστημα. Ε, σχεδόν υπαρξιακό. Γι' αυτό η πολιτική προσοχή θα στραφεί εκεί. Θα υπάρξουν και άλλες ευκαιρίες για να δοθεί, να δοθεί κατεύθυνση, ας πούμε, για αυτά τα θέματα, να ακούσουμε τις απόψεις του Κοινοβουλίου τους επόμενους μήνες, καθώς θα ξεκαθαρίζει ο ορίζοντας και η εικόνα. Ε, αυτή τη βδομάδα η Επίτροπος Μάστρομ θα πάει σε μια μικρή υπουργική ε, συνεδρίαση ε, στα περιθώρια των συζητήσεων του Νταβός. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Όντως, θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται και η στρατηγική σε σχέση με την Ινδία, τις ΗΠΑ και τους υπόλοιπους εταίρους μας και η Ευρωπαϊκή Ένωση σίγουρα μπορεί να παίξει το ρόλο της και να ακολουθήσει τη συγκεκριμένη της στρατηγική αλλά και να υποβάλει συγκεκριμένη πρόταση ώστε να πιέσει και τους υπόλοιπους να τηρήσουν, να παραμείνουν μάλλον στο πολυμερές σύστημα. Θα γίνει κάποια, θα έχουμε και άλλες ευκαιρίες για συζήτηση, όπως σας ανέφερα και, και νωρίτερα. Εμείς ως Κοινοβούλιο είναι καθήκον μας να εξετάσουμε πρώτα απ' όλα να δούμε την ε, κοινοβουλευτική ε, διάσκεψη. Θα υποβάλουμε σύντομα και ένα ε, έγγραφο για μεταρρυθμίσεις και θα πιέσουμε και τους συναδέλφους από άλλα κοινοβούλια να είναι πιο δραστήριοι. Έπειτα, θα θέλαμε να συζητήσουμε το μέλλον ε, της ε, γεωργίας ε, με τους επιτρόπους γιατί είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα πάντοτε στην ημερήσια διάταξη του ΠΟΕ. Ίσως με κάποιους άλλους ομιλητές και έπειτα αναφερθήκατε και στο, σε, στα σεμινάρια, η εργαστήρια με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες για το πώς δηλαδή θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε την εργασία εντός του ΠΟΕ. Να είναι δηλαδή αυτό κομμάτι της ημερήσιας μας διάταξης για φέτος. Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση λοιπόν για τα πορίσματα της 10ης Υπουργικής Διάσκεψης του ΠΟΕ. Πάμε στο σημείο 20, ε, ε, ετήσια έκθεση ε, σχετικά με την εφαρμογή της κοινής εμπορικής πολιτικής και η συγγετήρια είναι η κυρία Σαΐφη και της δίνω αμέσως το λόγο. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Σήμερα σας παρουσιάζω το σχέδιο έκθεσης που θέλω να παρουσιάσω σε σχέση με την κοινή εμπορική πολιτική. Πρόκειται για μια ανάλυση ε, της εμπορικής στρατηγικής ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βασίστηκα σε τέσσερα έγγραφα αναφορά. Στην ε, στρατηγική εμπόριο για όλους, το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2016 για την εμπορική στρατηγική, την έκθεση τη επιτροπή που δημοσιεύθηκε το περσμένο Σεπτέμβριο για την κατάσταση πρόοδου τη εμπορική στρατηγική δύο χρόνια μετά από την εφαρμογή τη και την έκθεση της ε, ε, Κομισιόν τη 9 η Νοεμβρίου για την εφαρμογή των Συμφωνιών Ελευθέρων Συναλλαγών. Η εφαρμογή τη εμπορική πολιτική συμπεριλαμβάνει διάφορα στοιχεία και συγκεκριμένα την πρόοδο των εμπορικών συμφωνιών, την παρακολούθηση τη εφαρμογή των νομοθετικών κειμένων και την ε, αξιολόγηση όλων όλων αυτών. Έχω υποβάλει, ε, μάλλον έχω μελετήσει τα έγγραφα αυτά και έχω υποβάλει τα πορίσματα και προς την Επιτροπή και κάποιες ερωτήσεις. Η αμοιβαιότητα και η εγγύηση για θεμητό ανταγωνισμό θα πρέπει να καθοδηγούν την εφαρμογή της εμπορικής πολιτικής της Ένωσης μέσω όχι μόνο των εμπορικών διαπραγματεύσεων αλλά και μέσω των εργαλείων που ε, ε, συστήνουμε θα πρέπει να αποτελεί ένα κεντρικό στοιχείο του μηνύματος που μεταφέρει το Κοινοβούλιο. Η Ένωση θα πρέπει να αντιδρά και να παρεμβαίνει άμεσα σε περίπτωση της λειτουργίας ή μη σεβασμού των εμπορικών δεσμεύσεων. Η Ένωση οφείλει να χρησιμοποιεί όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της και να ε, είναι ταχύτερη. Θα πρέπει να προτρέξουμε όσον αφορά την εφαρμογή των εμπορικών μας πολιτικών και να μεριμνήσουμε την καλή της εφαρμογή πριν να είναι αργά. Προ αυτή την κατεύθυνση ζητώ η εφαρμογή τη κοινή εμπορική πολιτική ε, να αποτελέσει αναπόσπαστο τμήμα τη εμπορική στρατηγική τη Ένωση και γι' αυτό το λόγο ζητώ οι ανθρώπινοι και οι οικονομικοί πόροι να αυξηθούν και να δημιουργηθεί μια ειδική ε, υπηρεσία μέσα στην Επιτροπή. Επανέρχομαι επίση στην πρώτη έκθεση τη Κομισιόν για την εφαρμογή των Συμφωνίων Ελευθέρων Συναλλαγών και ε, με ανησυχεί το γεγονό ότι οι Ευρωπαϊκέ επιχειρήσει δεν χρησιμοποιούν τις ε, εμπορικές προτιμήσεις που περιλαμβάνονται στις συμφωνίες ή Κομισιόν θα πρέπει να το διορθώσει αυτό και να αναπτύξει καλύτερη επικοινωνία και να συνοδεύει τι επιχειρήσει ώστε να μπορούν να εκμεταλλευτούν αυτέ τι συμφωνίε. Είναι επίση θεμελιώδου σημασία να συνεχίσουμε να, συστη... να συντάσσουμε ειδικά μέτρα για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Η έκθεση τη εφαρμογή για την εφαρμογή των συμφωνιών αφιερώνει ιδιαίτερο κομμάτι στι μικρομεσαίε, πράγμα που επιτρέπει καλύτερη ανάλυση και βελτίωση των, διατάξεων περί, ε, ε, περί μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Επίσης, η συνοδεία στις εξαγωγές θα πρέπει να αναπτυχθεί για τις μικρομεσαίες. Επανέρχομαι επίσης στα εργαλεία που επιτρέπουν στην εμπορική πολιτική να συμβάλλουν στην πρόθεση και την περάσπιση των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην ανάπτυξη μιας υπεύθυνη ε, διαχείρισης της αλυσίδας των αξιών. Το έχουμε ήδη συζητήσει στην πρώτη ανάλυση. Ε, ε, επιμένω στην σημασία να αναπτυχθεί η διαφάνεια και η πρόσβαση στις πληροφορίες, καθώς και να βελτιωθεί η ποιότητα των μελετών αντικτύπου. Ε, να δημοσιεύεται δε η διαπραγματευτική εντολή και πιο συγκεκριμένα να ενημερώνεται η εντολή αυτή κάθε πέντε χρόνια ώστε να μπορεί και να προσαρμόζεται. Καλό δε την Επιτροπή και τα κρατημένα να αναπτύξουν μια πραγματική ε, επικοινωνιακή στρατηγική γύρω από την εμπορική πολιτική και να συμπεριλάβουν εκεί περισσότερο τους ενδιαφερόμενους φορείς ώστε να λαμβάνουν τις πληροφορίες και τις απαντήσεις στις ερωτήσεις τους. Ε, αυτά θα έχω να πω για την ώρα, αν και υπάρχουν και άλλα στοιχεία στο σχέδιο έκθεσης και θα προσέξω πολύ τα σχόλια των συναδέλφων. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε και από τους εισελουστές η Καρολίνα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την πρόταση, αλλά νομίζω ότι Καλύτερα θα ήταν να τοποθετηθεί εκ μέρους μας Τζουντ. Εκπροσωπώ τον, τον, τον Τζουντ, ο οποίος θέλει να ευχαριστήσει την εισηγήτρια για το εξαιρετικό προσχέδιο της, το οποίο θέτει ένα πολύ καλό ε, πλαίσιο και για το περιεχόμενο και για την περίοδο. Αυτό είναι πολύ καλό, αν θέλουμε η έκθεση να είναι αποτελεσματική. Όσον αφορά τα θέματα που καλύπτει, χαιρόμαστε που ε, συμπεριλαμβάνονται πολλές από τις προτεραιότητες μας, ιδίως όσον αφορά την εφαρμογή των κεφαλαίων TST. Θα θέλαμε ωστόσο να υπερβούμε λίγο αυτά τα όρια και να κάνουμε συγκεκριμένες συστάσεις στην Κομισιόν. Θα υποβάλουμε και σχετικές τροπολογίες, κάποιες από τις οποίες θα βασίζονται και σε θέσεις που έχει λάβει και υιοθετήσει η Επιτροπή μας, αλλά και σε κάποιες νέες ιδέες. Για παράδειγμα, πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί καλύτερα το δίκτυο των ευρωπαϊκών αντιπροσωπιών. Το σχέδιο έκθεσης επίσης θέτει ένα θετικό πλαίσιο για την ε, αξιολόγηση από την πλευρά της Κομισιόν των συμφωνιών που έχουν συναυθεί. Θα μπορούσαμε για παράδειγμα επίσης όμως να ε, ασκήσουμε κριτική στο χαμηλό επίπεδο αξιοποίησης και χρήσης ε, των μέσων που έχουμε στη διάθεσή μας. Υπάρχουν ωστόσο και κάποια ζητήματα ποσοτικά και ποιοτικά που δεν ε, καλύπτονται επαρκώς ακόμη κατά τη γνώμη μας. Και γι' αυτό θα υποβάλουμε συγκεκριμένες πρωτοπολογίες που θα δίνουν συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές για το τι χρειάζεται ε, σε σχέση με την εφαρμογή των FTA. Και βεβαίως προσβλέπουμε στην καλή συνεργασία και στο συμβαστικό πνεύμα που θα επιδείξουμε όλοι και οι άλλοι σκιώδες. Ευχαριστώ. Κύριο από το ECR. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ε, ευχαριστήσω την εισηγήτριά μας για την έκθεσή της. Πιστεύουμε ότι έχει διατυπωθεί πολύ καλά και ως προς τη δομή της και ως προς το περιεχόμενό της. Αντικατοπρίζει τα γεωπολιτικά δεδομένα και υποστηρίζουμε τις περισσότερες από τις συστάσεις της. Έχουμε τρία ερωτήματα ή τρεις επιφυλάξεις αν θέλετε, που, ε, τις οποίες και θα αναπτύξουμε και σε τροπολογίες μας. Η μία αφορά την παράγραφο 20 που τονίζει την ανάγκη για αύξηση των ανθρώπινων και δημοσιονομικών πόρων σχετικά με την εφαρμογή των Συμφωνιών Ελευθερών Συναλλαγών. Είναι αλήθεια αυτό, ωστόσο το ίδιο ισχύει και για την φάση της διαπραγμάτευσης και της υπογραφής των ε, εμπορικών συμφωνιών. Και θέλουμε να τονιστεί αυτό. Αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, ε, βρισκόμαστε σε συζητήσεις με η Ιαπωνία Βιετνάμ και Σιγκαπούρη που βρίσκονται στο στάδιο της διαπραγμάτευση. Θα έπρεπε ήδη να έχουμε λάβει γνώση αυτών των εμπορικών συμφωνιών. Παρόλα αυτά ε, παρατηρούμε κάποιες καθυστερήσεις ε, και αυτό και πιστεύουμε ότι η Κομισιόν θα έπρεπε να έχει τους απαρκείς πόρους προκειμένου να ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έγκαιρα. Για την παράγραφο 4, τώρα δεύτερη επιφύλαξη, όσον αφορά την ανάγκη ε, ενίσχυσης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Προφανώς γνωρίζετε ότι ως CCR εμείς ε, διαφωνούμε με την ύπαρξη αυτού του ε, ταμείου. Έχουμε αντίθετη γνώμη. Δεν θεωρούμε ότι υπάρχει λόγος να υπάρχει ένα τέτοιο ταμείο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι' αυτό θα προτιμούσαμε μέτρα σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, τα οποία θα μπορούσαν και να προσαρμοστούν πολύ καλύτερα στις ανάγκες της κάθε περίπτωση. Τρίτον, θα θέλαμε να υπάρχουν περισσότερε αναφορέ στο ψηφιακό εμπόριο και τη σχετική στρατηγική που θα ακολουθήσουμε ω Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά ω προ τι επιφυλάξει μα, Γενικά όμω επαναλαμβάνω ότι ε, μας ικανοποιεί ε, το σχέδιο έκθεση. Σε αυτά τα τρία θέματα εμεί θα επιμένουμε. Κατά τα άλλα όμω βεβαίω προσβλέπουμε και στη συνεργασία με του άλλου σκιώδεις για να καταλήξουμε σε ένα θετικό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πολύ aber jetzt. Vielen Dank für den Vorschlag. Es handelt sich hier um einen sehr Κυρία Χάιντς, ευχαριστώ πολύ για την πρόταση. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική έκθεση που αφορά την εφαρμογή των ε, εμπορικών συμφωνιών. Γνωρίζουμε όλοι ότι τα πράγματα δεν εξελίσσονται πάντοτε κατευχήν. Γι' αυτό και χρειάζεται να βελτιωθούν οι διαδικασίε παρακολούθηση αλλά και αξιολόγηση εκ των υστέρων και αυτό πρέπει να τονίζεται στην έκθεσή μα ε, ω απέτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Για μένα είναι πολύ σημαντικό ε, να ε, τονίζεται ότι δεν αρκεί βεβαίως να συνάπτονται αυτές οι εμπορικές συμφωνίες μόνο, αλλά πρέπει να παρακολουθούνται ε, από κοντά και οι διαδικασίες εφαρμογής των εμπορικών συμφωνιών αυτών προκειμένου να μην υπάρχουν παραβιάσεις. Γι' αυτό το σκοπό βεβαίως απαιτείται και η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, της κοινωνία των πολιτών προκειμένου και αυτές να συμπεριλαμβάνονται στο μέλλον σε διαδικασίες ε, παρακολούθησης, αξιολόγησης. Επίσης, ε, οι κοινωνικοί εταίροι και η κοινωνία των πολιτών μπορούν να βοηθήσουν και με την υποβολή και την ανάδειξη και βέλτιση των πρακτικών. Επίσης, ε, νομίζουμε ότι θα πρέπει να προβλέπεται και ένας μηχανισμός επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση παραβιάσεων των εμπορικών συμφωνιών. Άρα, το δικό μας ζητούμενο είναι πώς θα συμμετέχουν περισσότερο οι κοινωνικοί εταίροι στη διαδικασία αυτή. Επίσης, σημαντικό για μας είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμμετέχει ε, ενεργότερα στη διαδικασία και μάλιστα από την αρχή, από την ε, έγκριση της εντολής έως και την υπογραφή της εκάστοτε συμφωνίας. Επίσης, ένα ακόμη θέμα που αφορά την φοροαποφυγή ε, εδώ νομίζω ότι χρειάζεται να γίνει και μια αναφορά στην καταπολέμηση της διαφοράς και την προστασία των πληροφοριοδοτών. Ένα άλλο θέμα που μας ενδιαφέρει και εμάς είναι το ζήτημα των ψηφιακών υπηρεσιών και εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι η διασυνοριακή ροή δεδομένων θα πρέπει να συμφωνεί με τους κανόνες προστασίας των προσωπικών δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για παράδειγμα θα μπορούσε ε, να υπάρχει μια οριζόντια ρήτρα σχετική για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στις, ε, στις ε, συμφωνίες. Κατά τα άλλα θα ήθελα να ευχαριστήσω βεβαίως την συγγήτρια για το έργο της και προσβλέπω και εγώ στη συνεργασία μαζί της. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ προσωπικά να αναφερθώ στην παράγραφο 22 που αφορά τον ρόλο των ενωσιακών ε, αντιπροσωπιών. Το ερώτημά μου προς την κυρία Άτσο είναι το εξή. Ποιο ρόλο επιτελεί η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης στη φάση της εφαρμογής των ε, συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών. Αίσθησή μου είναι ότι υπάρχει ακόμα μια προσέγγιση κατακαιρματισμένη. Ότι ε, η Γενική Διεύθυνση Εμπορίου ε, ασχολείται με τα οικονομικά ζητήματα και η Ευρωπαϊκή Εξωτερική, ε, Υπηρεσία Εξωτερική δράση ασχολείται με τα πολιτικά θέματα. Δεν υπάρχει μια ολοκληρωμένη δηλαδή στάση και προσέγγιση από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την εφαρμογή αυτών των εμπορικών συμφωνιών. Είναι η αίσθησή μου. Ε, δεν ξέρω αν έχω δίκιο, αλλά είναι η αίσθησή μου. Και δεύτερον, δεν υπάρχει κάποιο πρότυπο, κάποια τυποποιημένη διαδικασία σχετικά με την εφαρμογή των εμπορικών συμφωνιών. Υπάρχουν ε, στο, σε ολόκληρο τον πλανήτη αντιπροσωπείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ε, ασχολούνται ενεργά με την εφαρμογή των εμπορικών συμφωνιών, ενώ υπάρχουν και άλλες αντιπροσωπείες που απλώς παρακολουθούν τη διαδικασία αυτή. Μήπως θα έπρεπε λοιπόν να καταρτήσουμε συγκεκριμένες προδιαγραφές που θα διέπουν την εφαρμογή των εμπορικών συμφωνιών. Βεβαίως υπάρχει απέτηση η υποστήριξη των ε, αντιπροσωπιών στο έργο τους. Κάποιες πράγματι υποστηρίζονται και βοηθούνται κεντρικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, άλλως λιγότερο. Πώς μπορούμε λοιπόν να βελτιώσουμε, είναι το ερώτημα για μένα, των αντιπροσωπιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ολόκληρο τον κόσμο με σκοπό την καλύτερη εφαρμογή των εμπορικών συμφωνιών που έχουμε συνάψει με άλλες χώρες. Η εισηγήτρια έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Άκουσα πολλά σχόλια. Προκαταρτικά, να πω δύο λόγια για την έκθεση. Πριν μπω στην ουσία των ερωτήσεων για, την, ε, για το ρόλο των αντιπροσωπιών και το ρόλο των ε, συμφωνιών ελευθέρου εμπορίου. Καταρχάς, καλωσορίζουμε τις λεπτομέρειες που έχει βάλει στην εκθεσή του το ε- Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, στην έκθεση εφαρμογής της ε, Συμφωνίας των Συμφωνιών Ελευθέρου Εμπορίου. Ξέρετε πολύ καλά ότι εξετάζουμε όλες τις συμφωνίες ελευθερου εμπορίου υπό ελευθερου εμποριου που εφαρμογη και περιμένουμε προτάσεις και σχόλια από τα μέλη της Επιτροπής σας για το πώς θα ενισχύσουμε τι δουλειά μπορούμε να κάνουμε, για να ενισχύσουμε τη δουλειά που μπορούμε να κάνουμε. Για το ρόλο τώρα των αντιπροσωπιών. Έχουν σημαντικό ρόλο στη φάση εφαρμογής. Μπορούμε να μιλήσουμε για εκείνες τις αντιπροσωπίες όπου ασχολούνται με μία συμφωνία ελευθέρου εμπορίου που πρέπει να εφαρμοστεί π.χ. η αντιπροσωπεία στην ε, Σεούλ. Γιατί θα εφαρμόσουμε τη Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου ή μάλλον εφαρμόσουμε τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με την Κορέα εδώ και πέντε χρόνια. Και επομένω ε, έχει καλή εμπειρία η αντιπροσωπεία μα από εκεί. Ο βασικό ρόλο των αντιπροσωπιών είναι να φέρουν σε επαφή τα μέλη των πρεσβειών των κρατών μελών με τους επιχειρηματίες που βρίσκονται επί τόπου και να εντοπίσουν οποιαδήποτε εμπόδια ή οποιαδήποτε θέματα τέλος πάντων αφορούν την εφαρμογή μιας συμφωνίας ελευθέρου εμπορίου. Συχνά υπάρχει μια λεπτή γραμμή ανάμεσα στις δεσμεύσεις που, έχει αναλάβει, έχουμε αναλάβει μέσω των συμφωνίων ελευθερού εμπορίου σε σχέση με, τα, με τους φραγμούς που υπάρχουν για την πρόσβαση στην αγορά. Ε, η υπηρεσία εξωτερικής δράσης και οι αντιπροσωπείες Ευρωπαϊκής Ένωσης παίζουν σημαντικό ρόλο εδώ. Γιατί παρακολουθούν μεταξύ άλλων την εφαρμογή της συμφωνίας στα διάφορα κεφάλαια, κεφάλαιο προς κεφάλαιο, σε διάφορους τομείς. Ξανά θα μπω στο παράδειγμα της Κορέας. Έχουμε παραδείγματος χάρη διάφορα κεφάλαια που αφορούν διάφορους τομείς. Εντοπίζοντας τους φραγμούς και θέτοντας το θέμα αυτό στις κανονιστικές επιτροπές και στις ομάδες εργασίας, όπου συζητούνται τα θέματα εφαρμογής με τους εταίρους, ε, γίνεται μια πολύ σημαντική δουλειά. Έχουμε πολυάριθμες ε, συμφωνίες ελευθερού εμπορίου και αυξάνονται όλο και περισσότερο. Ακριβώς γι' αυτό η ιεράρχηση για την Κομισιόν και τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου είναι πολύ σημαντική ε, όπως και για την υπηρεσία εξωτερική δράση βεβαίως. Είναι σημαντικό λοιπόν να υπάρξει μια ιεράρχηση. Ευχαριστώ. Κυρία. Η κυρία Σάιφη τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους ε, για τις παρεμβάσεις τους. Διαπιστώνω ότι υπάρχει μια μεγάλη συνένεση για τους ε, βασικούς προσανατολισμούς ε, στις συζητήσεις της Επιτροπής μας. Συμφωνώ με την παρατήρηση που κάνετε για την αδυναμία ορισμένων αντιπροσωπιών και το θέμα της εφαρμογής. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να το παρακολουθούμε. Άκουσα όλες τις παρεμβάσεις. Ε, να πω κάτι για το ψηφιακό εμπόριο. Ίσως θα έπρεπε να ξαναδούμε και να ενισχύσουμε το θέμα του ψηφιακού εμπορίου. Προσοχή λοιπόν, προσοχή στις τροπολογίες που θα κατεθούν και αυτό το θέμα και είμαι έτοιμη να συνεργαστώ με τους κοιόδης εισηγητές. Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε. Είναι μια σημαντική έκθεση αυτή. Και καλωσορίζουμε την δουλειά που έκανε η συγγητριά μας. προθεσμία για τις τροπολογίες 30 Ιανουαρίου. Τόσο Σονούπο δηλαδή. Τι, τι ώρα να βάλουμε, 10 η ώρα ή 12, 12 η ώρα. Πολύ ωραία. Μία εβδομάδα έχουμε για τις τροπολογίες εδώ στην Ίντα και θα συζητήσουμε μετά τις τροπολογίες στις 19 και 20 Φεβρουαρίου. Σας ευχαριστώ. Σημείο 21. Ερμηνεία και εφαρμογή της Διοργανικής Συμφωνίας για την βελτίωση του νομοθετικού έργου. Ο κύριος Μπέντσεν είναι ο εισηγητής μας. Δεν είναι εδώ, αλλά θα έρθει όπου να είναι. Κάνουμε ένα δίλεπτο διάλειμμα. Ελπίζουμε στο μεταξύ να έχει έρθει ο εισηγητής μας. Ευχαριστώ. <laughs> Okay, so I reopen the session and we... Αρχίζουμε. Πάμε στο 21. για την εφαρμογή και ερμηνεία της Διοργανικής Συμφωνίας για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Εφαρμόζω ε, και παρακολουθώ τη ρήτρα εφαρμογής. Είμαι συνεισηγητής για αυτό το θέμα, για τις προφορίες για τις διεθνείς συμφωνίες, εγώ και ο συνάδελφος ε, διαπραγματευόμαστε με το Συμβούλιο. Εδώ και 1,5 χρόνο. Και δεν είναι εύκολο να διαπραγματευτεί κανείς με το Συμβούλιο ή μάλλον με την νομική υπηρεσία του Συμβουλίου για να υπάρξει μια συμφωνία που θα αντικατοπτρίζει τις σαφείς προϋποθέσεις και ανάγκες της Συμφωνίας της Λισαβόνας. Θα πρέπει να, έχουμε, να είμαστε ισότιμοι με το Συμβούλιο, θα πρέπει να έχουμε όλα τα στοιχεία των διαπραγματεύσεων των εμπορικών, από την, ε, τον προβληματισμό, την εντολή, την ε, περίοδο διαπραγμάτευσης μέχρι την εφαρμογή. γιατί θέλουμε να ξέρουμε τι γίνεται στο, στην εμπορική πολιτική. Έχουμε ακούσει τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι η Γενική Διεύθυνση Εμπορίου θα μας δίνει όλες τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της. Αλλά δεν είναι αυτή όλη η εικόνα. Και επιπλέον, ε, υπάρχουν πολλές ε, συμφωνίες διεθνείς συμφωνίες που αφορούν διάφορες κοινοβουλευτικές επιτροπές. Παραδείγματος χάρη η Επιτροπή Αλίας ε, έχει τις αλληλευτικές συμφωνίες. Δεν έχουμε όλοι τις ίδιες πληροφορίες για τις συμφωνίες αυτές τις διεθνείς. Δεύτερο βασικό στοιχείο στη διαπραγμάτευση είναι είναι ότι το Συμβούλιο κάνει προσωρινή εφαρμογή μιας συμφωνίας που ανησυχούσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εδώ η Επίτροπος Μάστρομ είχε δεσμευτεί ότι δεν θα γίνει αυτό στον τομέα του εμπορίου, έχει γίνει σε άλλο τομέα προσωρινή εφαρμογή. Αλλά το εμπόριο είναι μόνο ένα τμήμα της εξίσωσης. Έχουμε διάφορες συμφωνίες και είναι εντελώς ασαφές εάν οι θέσεις και οι απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορούν να επηρεάσουν καθόλου τη διαδικασία σε διάφορες κοινοβουλευτικέ επιτροπές σκέφτονται τώρα να μην προχωρήσουν στην διαδικασία του Συμβουλίου, ούτως ώστε να μην υπάρξει καμία προσωρινή εφαρμογή. Γιατί το κοινοβούλιο θα απόσχει, δεν θα, θα παίξει αυτό το παιχνίδι, ας πούμε. Είναι περίεργη και επικίνδυνη αυτή η στρατηγική, γιατί μπορεί να είναι επιζήμια για τρίτα μέρη. Και εμείς λοιπόν δεν είμαστε πολύ υπέρ αυτής της διαδικασίας του να μην παίξουμε καθόλου σε αυτό το παιχνίδι. Για να αποφύγουμε αυτή τη διαδικασία, ο κ. Μπροκ και εγώ προτείναμε στη διάσκεψη των Προέδρων την περασμένη εβδομάδα να προετοιμάσουμε ε, ένα κείμενο προς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ε, οι πολιτικές ομάδες και το Κοινοβούλιο συμφώνησε με την πρόταση αυτή και ο Πρόεδρος έγραψε μία επιστολή στη νομική μας υπηρεσία για να προετοιμάσει ε, ένα κείμενο νομικό, δεσμευτικό και ελπίζω αυτό να φέρει μια νέα πνοή στο Συμβούλιο και να επηρεάσει και τη διαπραγμάτευση που έχουμε που θα λάβει χώρα Είμαστε έτοιμοι να πάμε στο δικαστήριο εάν δεν έχουμε αποδεκτό αποτέλεσμα από το Συμβούλιο τους επόμενους μήνες. Φυσικά, αν βγει μια τέτοια εικόνα, ας πούμε, ότι τα θεσμικά όργανα καυγαδίζουν, αυτό δεν είναι μια ελκυστική εικόνα που προβάλλουμε, αλλά χρειαζόμαστε ίση μεταχείριση, περισσότερες πληροφορίες, περισσότερη διαφάνεια, για να παίξουμε το ρόλο μας ως κοινοβούλιο και να ελέγξουμε την όλη διαδικασία δηλαδή, των διαπραγματεύσεων για συμφωνίες σε διεθνές επίπεδο. Αυτή ήταν μια σύντομη παρουσίαση τι έχουμε κάνει, του τι έχουμε κάνει και τώρα θα δώσω το λόγο στον εισηγητή μας. so much, uh, uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τις πληροφορίες για τις άμεσες διαπραγματεύσεις που γίνονται σε αυτόν τον τομέα. Ήδη έχουμε συζητηθεί. Στις 4 Δεκεμβρίου 2017 είχαμε συζήτηση όπου τα συζητήσαμε τα προβλήματα το σχέδιο τώρα γνωμοδότησης ε, είναι έτοιμο. Ξέρουμε ότι η προθεσμία για υποβολή τραπολογιών 26 Ιανουαρίου, την επόμενη ε, Παρασκευή. Και ε, το συζητήσαμε αυτό και πέρυσι, όπου είδαμε ότι υπήρχε πρόβλημα με την υπηρεσία εξωτερικής δράσης όπου μας αγνοούν. Και πριν δώσει τη συνέντευξή του το Κοινοβούλιο, ε, εφαρμόζουν προσωρινά τις συμφωνίες. Το συζητήσαμε αυτό το θέμα. Ότι θα πρέπει καθ' όλη τη διάρκεια διαπραγμάτευσης μιας διεθνούς συμφωνίας να ενημερώνεται το Κοινοβούλιο από από τη φάση της διαπραγματευτικής εντολής μέχρι τέλους. Τα βάλα αυτά στο κείμενό μου. Τα έχουμε ξανασυζητήσει. Οι περισσότεροι από εμά ε, συμφωνούμε. Προσβλέπω λοιπόν να ακούσω τις ε, προτάσεις για τη βελτίωση του κειμένου από τους συναδέλφους. Δεν θα επαναλάβω όλα τα προβλήματα που είχαμε. Τα ανέφερε και ο πρόεδρος εξάλλου. Ακούσαμε τι μας είχε πει στο παρελθόν η Επίτροπος Μάρστρομ. Θέλουμε καλύτερη συμπεριφορά στο μέλλον. Αυτό βάζουμε και σε αυτή την ε, γνωμοδότηση λοιπόν. Ακριβώς αυτές τις ε, απόψεις. Αυτά εν συντομία. Ευχαριστώ. Και εγώ ω σκιώδη υποστηρίζω την γνωμοδότηση αυτή πλήρω. και κάποιες φορές πραγματικά η συμπεριφορά του Συμβουλίου είναι απίστευτη. Εμείς πάντοτε ζητούμε να συμμετέχουμε καταρχάς στην, ε, στην ζητούμε να υπάρξει εντολή και να υπάρξει και δημοσίευση αυτής της εντολής. Πολλές φορές η απάντηση σε αυτό είναι ότι βρισκόμαστε στο μέσο της διαπραγμάτευσης βάσει του άρθρου 40 και θα περιμένουμε με τη για τη δημοσίευση έως ότι ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση. Είναι τρελό. Έχουμε δικαίωμα ενημέρωσης. Είναι παράνομο αυτό που κάνει το Συμβούλιο. Ελπίζω λοιπόν η γνωμοδότηση αυτή να ασκήσει πίεση Κύριε Σόλτς, ευχαριστώ τον εισηγητή το, για τις εισαγωγικές του παρατηρήσεις συμφωνώ και εγώ ότι πρέπει να αγωνιστούμε μέχρι τέλους. Και αν χρειαστεί να προσφύγουμε μέχρι και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Και να υπερασπιστούμε το δικαίωμά μας να συμμετέχουμε στην ε, κατάρτιση των εντολών. Ε, Συμφωνώ επίση ότι θα πρέπει να καλύπτεται στη γνωμοδότησή μας και το ζήτημα της μελέτη αντικτύπου. Για παράδειγμα, το έχουμε ξανασυζητήσει το θέμα αυτό, ε, την μελέτη του Ολιβιέ Ντισκούτα, που αφορούσε τα ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο των ε, συμφωνιών ελευθερών συναλλαγών αρκεί η διαφάνεια από μόνη της ή θα πρέπει να υπάρχουν και συγκεκριμένες διατάξεις και ρήτρε σε συμφωνίες αυτές για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ζητούμε λοιπόν από την Κομισιόν να προβλέπει μηχανισμούς, εργαλεία για την ε, ε, επιβολή των όσων προβλέπονται. Ωστόσο, δεν έχουμε ε, επαρκή εργαλεία για να παρακολουθούμε την πρόοδο σε αυτό το θέμα. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτές οι ε, θέσεις θα πρέπει να διέπουν και την μελλοντική μας ε, κανονιστική συνεργασία. Κάτι που υπερβαίνει βεβαίως και τις αρμοδιότητες Επιτροπής ΙΝΤΑ. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε μια συμφωνία η οποία θα καλύπτει και τις εξωτερικές δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα διέπει εν γέννη τις δραστηριότητες και άλλων επιτροπών και σε άλλους τομείς. Επίσης, χρειαζόμαστε διαφάνεια σχετικά με τις δράσεις που αναλαμβάνει η Κομισιόν και άλλα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι γίνεται δηλαδή σε διάφορου διεθνεί οργανισμού, όπω είναι ο Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Και βεβαίω υπάρχουν και οι, ε, οι ομάδες που έχει συστήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και παρακολουθούν τα θέματα αυτά, αλλά χρειάζεται να υπάρχει μια μόνιμη δομή ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων για να μπορούμε να ενημερωνόμαστε για το τι κάνει σε κάθε στάδιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ζητεί κάποιο άλλο το λόγο. Όχι. Θα ήθελα λοιπόν να δώσω το λόγο τότε στην Κομισιόν. Η κυρία Ιωάννα Λέσουκ έχει το λόγο. Ναι, γεια σας κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ θα ήθελα να θυμίσω ότι έχουμε κάνει μια πολιτική συνεδρίαση στις 12 Δεκεμβρίου όσον αφορά την ε, πολιτική αξιολόγηση για την καλύτερη νομοθεσία καθώς ε, και ε, εκεί συμμετείχαν τα τρία θεσμικά όργανα και αναγνωρίστηκε κοινά η κοινή δέσμευση το άρθρο 50 της συμφωνίας και είναι κάτι που θα γίνεται ετήσια ε, όσον αφορά τις πρακτικές ρυθμίσεις για τις διεθνείς ε, συμφωνίες, ελπίζουμε ε, για επιτυχή έκφαση. Ευχαριστώ. Okay, so you really happy with the West? Ωραία. Ε, για το άρθρο 40 ε, περιμένουμε, γιατί το υπόλοιπο είμαστε ικανοποιημένοι. Εισηγητής μας και πάλι. Thank you so much for, for, for the... Σας ευχαριστώ πολύ για τα σχόλια και ευχαριστώ για τα σχόλια και θα δούμε ποια θέση θα είναι οι τροπολογίες και μετά θα το ξανασυντήσουμε. Πολύ ωραία. Προθεσμία είναι 26 Ιανουαρίου το μεσημέρι και το Μάρτιο θα ε, ψηφίσουμε στην Επιτροπή. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχουμε λίγο περισσότερο χρόνο για μεσημεριανό διάλειμμα, αλλά θέλω να σας θυμίσω ότι η ε, κρόαση θα, ξεκινήσει στις 2.30. Ακριβώς. Καλή σας όρεξη.